So, good morning, dear colleagues. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Είναι 9 και 10 ήδη. Και όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος μας, ο κύριος Λάγκε, Ο πρόεδρος σήμερα απουσιάζει γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, στην περιφέρειά του, επομένως θα προεδρεύω εγώ στη θέση του. Ε, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Δεν έχω κάποιες ανακοινώσεις, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθύς με το σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την επέκταση των διατάξεων ε, της ε, Συμφωνίας ε, Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με το Ουσβεκιστάν στον τομέα της κλωστοφαντουργίας. Έχουμε μία ώρα για αυτή τη συζήτηση. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους, με η συγγήτρια για το θέμα αυτό είναι η κυρία Μαρία Ρένα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και πρέπει να συζητήσουμε το γεγονός ότι το πρωτόκολλο για την κροστοϊφαντουργία δεν έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του ε, ε, Κοινοβουλίου και έχουμε μια προσωρινή έκθεση για το Ουσβεκιστάν. Ολομέλεια ακολούθησε την πρόταση και από τότε έχουμε τακτικέ συναντήσεις με του ενδιαφερομένους για να δούμε τι ε, πρόοδο έχει επιτελεστεί στο Ουσμπεκιστάν. Σήμερα η συγγήτρια η κυρία Ρένα οργανώνει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τη Διεθνή Οργάνωση εργασία. Έχουμε εδώ ε, προσκεκλημένους επιρρογνώμονε. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χάιντ ε, Κόλλαρ. Ο κύριο Κόλλαρ είναι περιφερειακό διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στη Διεθνή Οργάνωση εργασία η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας παρακολουθεί την ε, ε, συγκομιδή Βάμβακος από το 2013 στο Ουσμπεκιστέν και θα ε, γίνει η παρακολούθηση και φέτος και θα μας ενημερώσει για το κατά πόσο γίνεται σεβαστές οι συμβάσεις της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία στο Ουσμπεκιστάν. Έχετε το λόγο για 10, το πολύ 15 λεπτά. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά για μένα να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας εκ μέρους ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. θα σα παρουσιάσω μια εικόνα των πρόσφατων εξελίξεων στη συνεργασία με το Ουσμπεκιστάν και τη Διεθνή Οργάνωση εργασία, καθώ και τα προκαταρκτικά μα ε, στοιχεία για την παιδική και καταναγκαστική εργασία. Καταρχά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή σα για την υποστήριξη του ε, έργου του γραφείου μα στο Ουσμπεκιστάν, βάσει και του ψηφίσματος τη 15 5η Δεκεμβρίου του 2011. Έχουμε δύο τεχνικά προγράμματα συνεργασίας στο Ουσμπεκιστάν. Το ένα συνδράμει ε, το ε, συνολικό πρόγραμμα αξιοπρεπούς εργασίας και το άλλο είναι τμήμα της συνεργασίας μας με την Παγκόσμια Τράπεζα και διασφαλίζει παρακολούθηση και αξιολόγηση της συγκομιδής Βάμβακος. Και τα δύο προγράμματα εξετάζουν ε, τι δράση έχει ανακοινωθεί και τι έχει εφαρμοστεί από πλευράς κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αυτή η τριμερή συνεργασία μας έχει οδηγήσει σε αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων, κυρίως ε, την παιδική εργασία. Ήταν το βασικό ε, στοιχείο πριν από τρία χρόνια ε, για τη συνεργασία που αναπτύσσεται τώρα. Ω τμήμα αυτής της διαδικασίας, τα συνδικάτα του Ουσβεκιστάν και το Εμπορικό Επιμελητήριο έχουν ε, δημιουργήσει και ενισχύσει δεσμούς ε, με διεθνείς οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και ε, πλέον ο κλωστό εφαντουργικό τομέας του Ουσβεκιστάν συμμετέχει στη Διεθνή Οργάνωση Εργοδοτών. Το Συνδικάτο του Ουσβεκιστάν συμμετέχει στην Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων αυτή η σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του Ουσβεκιστάν, ήταν επίσης και κινητήριος μοχλός για αυτή τη συνεργασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το, η Διεθνή Ομοσπονδία Συνδικάτων βοηθά το Σμπεκιστάν για να δημιουργήσουν τη λεγόμενη νομική κλινική, legal clinic, σε περίπτωση που υπάρχουν ε, νομικά προσκόμματα για την ε, παιδική και καταναγκαστική εργασία γίνεται ένας ε, παραδοσιακός ε, γύρος, πρώτης, γύρος τραπέζης πρώτης συγκομιδής ε, στην Τασκένδη και εκεί συμμετέχει η Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Παγκόσμια Τράπεζα και πριν από τέσσερις εβδομάδες διεξήφθη ο τελευταίος γύρος και θα σας πω κάποια στοιχεία. Καταρχάς, το πρόγραμμα συνεργασίας για την αξιοπρεπή εργασία που είναι το πρώτο στην Κεντρική Ασία θα ανανεωθεί από το τέλος του έτους. Δεύτερον, έχουν γίνει συγκεκριμένε εργασίε για να κατανοήσουμε καλύτερα τι προβλήματα υπάρχουν με την ε, πρόσληψη εργατικού δυναμικού για τις γεωργικές εργασίες και κυρίως ε, η μεγάλη κλίμακας οργάνωση της συγκομιδής Βάμβακος και επίσης ε, τα όσα ξεκίνησαν το 2013 για την παρακολούθηση της συγκομιδής Βάμβακος για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την παιδική εργασία και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις για την αξιοπρεπή εργασία. Κυρίως επικεντρωνόμαστε στην ε, στον περιορισμό της χρήσης καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας. Το πρόγραμμα της χώρας για την αξιοπρεπή εργασία είναι το βασικό στοιχείο που έχουμε ε, χρησιμοποιήσει για τις δραστηριότητες μας. Ε, κυρίως έχουμε σταθεί στη γεωργία και στην παιδική εργασία, σε νομοθετικά θέματα με τις σχετικές συμβάσεις και τριμερή συνεργασία θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία δυνατοτήτων για τους ε, εργοδότες και τους εργαζομένους και επίσης ξεκινήσαμε τώρα να καταρτίζουμε το επόμενο πρόγραμμα αξιοπρεπούς εργασίας για να επικεντρωθούμε και σε τομείς όπου μπορούμε να έχουμε και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε επιτυχία έχει επιτελεστεί για την ε, εξάλληψη της παιδικής εργασίας και την βελτίωση των ε, διαδικασιών πρόσληψης, ε, κυρίως θέλουμε να οδηγήσει σε βιώσιμα κατάλληλα μέτρα για την αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ικανότητες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρίως σε επίπεδο επαρχίας και σε τοπικό επίπεδο. Στο επόμενο στάδιο θα εξετάσουμε λοιπόν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες προκύπτουν από τον εξυγχρονισμό της ουσμπεκικής οικονομίας και κυρίως, αλλά όχι μόνο, τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Υπάρχουν επίσης θέματα ευρύτερα που αφορούν ε, πολιτική απασχόληση, ασφάλεια στο χώρο της εργασίας και ε, υγεία στον χώρο της εργασίας και επιθεώρηση εργασίας. Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε και με την Παγκόσμια Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα έχει καταρτήσει μια έκθεση που επισημαίνει κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξει το Ουσβεκιστάν. Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε τον Ιανουάριο φέτο ένα πρόγραμμα δράση για να βελτιώσει τι συνθήκε εργασία και την κοινωνική προστασία και ασφάλιση ε, στον τομέα τη γεωργία και αυτό συζητήθηκε με το Διεθνέ Γραφείο Εργασία πριν από την έγκρισή του. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία στα οποία και η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Γραφείο Εργασία πρέπει να συνεισφέρουν. Τώρα να περάσω στην ε, συνεχή έρευνα των συνθηκών πρόσληψης και εργασίας στην Γεωργία, κυρίως στη συγκομιδή Βάμβακος. Πέρσι παρουσιάσαμε μια ποιοτική ανάλυση που ανέλυε τα διάφορα στοιχεία τα οποία κυριαρχούν σε αυτό το τομέα και αυτή η ανάλυση τώρα ε, συμπληρώνεται από μια ποσοτική μελέτη. Τα στοιχεία αυτής της έρευνας αξιολογούν την κατάσταση και το 2014 και το 2015, ακόμα βέβαια τα ελέγχουμε και ε, η έρευνα διεξήχθη ως ε, έρευνα στα νοικοκυριά. Είχαμε 10.000 απαντήσεις και πλέον και πέρσι και φέτος και έχουμε κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα τα οποία παρουσιάστηκαν προς το παρόν, κυρίως για να βοηθήσουμε να... Ε, γνωστοποιηθούν κάποια θέματα για την παρούσα οικονομική χρονιά. Επίσης, ε, δώσαμε και τα στοιχεία στους Ουσμπέκους εταίρους μας, ε, ε, όπως σας είπα, στο γύρο τραπέζης που έγινε στην Τασκένδη πρώτη συγκομιδής. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα. Γύρω στους δύο μήνες διαρκεί η περίοδος συγκομιδής ε, και συμμετέχουν χιλιάδες εργαζόμενοι, πολλοί συμμετέχουν ε, θελοντικά. Κάποιοι όμως εξ αυτών μπορεί να διστάζουν, και, αλλά δεν μπορούν να αντισταθούν στις κοινωνικές πιέσεις από τους ομολόγους τους και ε, ορισμένες φορές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκομιδή. Βάσει των στοιχείων μας, η μεγάλη πλειονότητα συμμετέχει εθελοντικά όταν τους καλούν να ε, συλλέξουν βαμβάκι. Αυτές οι δραστηριότητες είναι απλώς ε, μια ε, δυνατότητα για επιπλέον εισόδημα. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους, από ό,τι φαίνεται, ότι ο ο αριθμός των ανθρώπων που ένιωσαν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν λόγω κοινωνικών πιέσεων μειώθηκε όσον αφορά αυτούς που ε, συλλέγουν βαμβάκι χωρίς τη θέλησή τους, ε, ε, φαίνεται ότι το βασικό στοιχείο είναι η απέτηση να πληρωθεί κάποιος άλλος για να κάνει τη δουλειά αυτή. Ένα από τα συμπεράσματα είναι να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος καταναγκαστικής εργασίας, διευκρινίζοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να υποχρεωμένος να πληρώσει ή να συλλέξει βαμβάκι αν δεν το επιθυμεί. Από τα ευρήματά μας ε, διαπιστώνουμε επίσης ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αρνούνται να συμμετέχουν έχει αυξηθεί ουσιαστικά. Μεταξύ του 2004 και του 2015 εκτιμούμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αρνούνται από 644.000 ανέβηκε στο 1 εκατομμύριο ε, άτομα. Και οι περισσότεροι εξ αυτών που αρνήθηκαν να συμμετέχουν δεν είχαν αρνητικές συνέπειες ή κάποια τιμωρία. Συνήθως είναι ε, η υποχρέωση να πληρώσουν κάποιον άλλον για να κάνει τη δουλειά αυτή αντί αυτών. Ε, αυτός οι πληρωμές που ζητούνται ως υποκατάστατο θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ε, σημείο εστίασης για την ε, διεθνή εκστρατεία η οποία στοχεύει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η εκστρατεία για εθελοντική συμμετοχή είχε θετικές συνέπειες ε, στο διάστημα 2014-2015. Επίσης, από την έρευνα επισημαίνεται ότι η ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν ε, εθελοντικά είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που δεν θέλουν και έχουν δισταγμούς και επίσης ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο εξυγχρονισμός της γεωργίας ε, θα σέβεται και ε, βασικές αρχές εργασίας. Από την έρευνά μας ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι λένε ότι θέλουν ούτως ή άλλως στο μέλλον να συμμετέχουν σε συνδρομητή βάμβακος λόγω του επιπλέον εισοδήματος. Πάνω από ένα εκατομμύριο λένε ότι θα ε, ε, συμμετείχαν αν υπήρχαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερη πληρωμή. Η παραγωγικότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν εθελοντικά φυσικά είναι μεγαλύτερη από αυτούς που συμμετέχουν καταναγκαστικά και βάσει των εκτιμήσεών μας η παραγωγικότητα μπορεί να είναι και 30% υψηλότερη. Άρα η όλη συγκομιδή θα μπορούσε να γίνεται με ανθρώπους που εργάζονται εθελοντικά ε, βάσει των προϋποθέσεων που μόλις σας επεσήμενα. Οι εταίροι μα στο Ουσμπεκιστάν ζήτησαν από το Διεθνέ Γραφείο Εργασίας να κάνει συστάσεις για περαιτέρω δράσεις βάσει της ποσοτικής έρευνας. Οι συστάσεις μας ε, είναι οι εξή. Οι αρχές πρόσληψης θα πρέπει να γνωρίζουν πώς γίνεται η πρόσληψη και ε, να γνωρίζουν και οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους να αρνηθούν να συλλέξουν βαμβάκι. Η εκστρατεία θα πρέπει να είναι πολύ καλά στοχευμένη και να είναι γενικότερη. Η αμοιβή και οι συνθήκες εργασίας θα πρέπει να είναι υψηλότερες. Και επίσης ε, προτείνουμε τα μέτρα για την εθελοντική πρόσληψη να ισχύουν για όλη την προσωρινή γεωργική εργασία και για την συγκομιδή βάμβακος εξετάζουμε το ενδεχόμενο να εφαρμόσουμε πιλωτικά προγράμματα των συστάσεων αυτών σε κάποιε περιοχέ. Και τέλο θα ήθελα να σα πω κάτι για την παρακολούθηση. Η πρώτη παρακολούθηση τη συγκομιδή Βάμβακο έγινε πριν από τρία χρόνια με στόχο κυρίω την παιδική εργασία. Η έκθεση του 2015 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, διαπιστώνει ότι η παιδική εργασία δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα σε γενικές γραμμές και μάλιστα θεωρείται και κοινωνικά απαράδεκτη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις παιδικής εργασίας και σίγουρα δεν θα πρέπει ε, να καθησυχαζόμαστε. Αλλά παρά το γεγονός ότι έχει εξαλειφθεί πλέον η παιδική εργασία, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις και πρέπει να τις καταπολεμήσουμε και αυτές. Η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστέν τα τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει σημαντικές δεσμεύσεις ε, και προς τις δύο κατευθύνσεις και για την εξάλληψη της παιδικής εργασίας και να διαπιστώσει ότι ε, θα υπάρχουν πρακτικές πρόσληψεις οι οποίες θα ε, αποτελούν κίνητρο για εθελοντική εργασία κυρίως βελτίωση της πρόσληψης και των συνθηκών εργασίας και φέτος θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς μεταφράζονται οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν σε πράξη. Κυρίως δηλαδή θέλουμε να δούμε συστημικά ζητήματα πρόσληψη. Όπω συζητήσαμε με τους εταίρου μας στο Ουσβεκιστάν, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα γίνονται από κοινού και πριν και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου και περιλαμβάνει και τη συγκομιδή που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες. Θα γίνουν επισκέψεις φοιτίες βάμβακα και ε, θα δούμε και οργανώσεις εργασίας στις αντίστοιχες περιοχές. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε περαιτέρω δράση σε διάφορα επίπεδα δηλαδή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι βασικοί στόχοι αυτών των εργασιών γίνονται σεβαστοί και ενισχύονται περαιτέρω. Είμαι πεπισμένος ότι και η εταίροι μας στο Ουσβεκιστάν και η διεθνής κοινότητα χρειάζονται τις ε, αξιολογήσεις μας για το πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας και πώς μπορεί να εξυγχρονιστεί περαιτέρω. Εμείς εξετάζουμε ε, εις βάθος τα θέματα, βλέπουμε τι δράση χρειάζεται για τις γεωργικές εργασίες και για όλη τη μορφή ε, εργασίας στο Ουσμπεκιστάν, ώστε να γίνεται με αξιοπρεπείς συνθήκες θα ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι ο Διεθνής, το Διεθνέ Γραφείο Εργασία θεωρεί ότι έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδο στο Ουσβεκιστάν τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι ε, κάτι το οποίο είναι εξελίξη. Θα χρειαστεί δουλειά και υποστήριξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κυρίως ως προς το θέμα της παιδικής εργασίας και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους η κυβέρνηση και η κοινωνική εταίρες στο Ουσβεκιστάν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Uh, thank Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόλεβαν. Σίγουρα οι ευρωβουλευτές θα έχουν ε, αρκετές ερωτήσεις για σας και για τους συναδέλφους σας. Τώρα, η Μαρία Ρένα. Θα δώσω το λόγο δηλαδή στα μέλη της Επιτροπής μας και πρώτα η Μαρία Ρένα, η συγκήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση γνωστή στην Επιτροπή μας γιατί αποτελεί μέρος της Συμφωνίας εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας ήδη την προηγούμενη και το 2011 είχαν διατυπωθεί διάφορες συστάσεις. Το πρωτόκολλο για την εφαντουργία επιτρέπει να συμπεριλάβουμε στην Συμφωνία εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας του 1999 και την κλωστεφαντουργία. Είχαν γίνει συναντήσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, με κυβερνητικούς και είχαμε δημιουργήσει εμείς διάφορες ομάδες ελέγχου. Η τελευταία είναι του Μαρτίου του 2016, όπου ήταν και συνδικάτα από το Ουσβεκιστάν παρόντες και ΔΟΕ και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δεκέμβριο του 2011 είχαμε διατυπώσει, όπως σας είπα, συστάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ουσβεκιστάν, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι εδώ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε εταιρική σχέση με την κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν αλλά και με τα συνδικάτα του Ουσβεκιστάν προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση όσον αφορά την καταδικαστική εργασία και την παιδική εργασία και το ακούσαμε και σήμερα ότι συμπεριλήφθηκε και το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα διάφορα δείγματα που μας φτάνουν και από τον ΔΟΕ και από τα συνδικάτα στο Ουσβικιστάν που συμμετέχουν ως παρατηρητές στα ευρωπαϊκά συνδικάτα Αυτές οι ενδείξεις λοιπόν, τα δείγματα είναι θετικά για να προχωρήσουμε. Επίσης δεσμευτήκαμε να καταλήξουμε σε απόφαση μέσα στους επόμενους μήνες για αυτό το θέμα. Προσοχή, μια πολιτική κατάσταση στο Σπεκιστάν σήμερα βρίσκεται υπό αλλαγές, οπότε την απόφασή μας πρέπει να τη θέσουμε και στο σημερινό πλαίσιο. να προχωρήσουμε στην ε, επικύρωση του πρωτοκόλου με ε, επισυνάπτοντας όμως και ένα κείμενο με επιχειρήματα σχετικά με την απόφασή μας. Όντως ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνομιλητές για το πολύ σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί. Σημειώνω ότι είναι μία από τις χώρες που είναι πιο ανοιχτές, που δέχεται εδώ και πάνω από τρία χρόνια σήμερα παρατηρητές από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό και γι' αυτό θέλουμε αυτή τη συμφωνία με το Βικιστάν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για το έργο τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την εισηγήτρια, τώρα οι πολιτικές ομάδες. ΕΛΚ πρώτα. Ντάνιελ, έχεις το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, από πλευρά τη Κιόδου εισηγήτρια που έχει ασθενήσει και αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παραστεί, Πρώτον μου ζήτησε να χαιρετήσω θερμά και να παρακαλέσω το πρωτόκολλο παρόλες τις αδιαμφισβήτες δυσκολίες να το εγκρίνουμε. Και δίκαια στο ψήφισμα είχαμε ζητήσει ότι αναμένουμε χειροπιαστές βελτιώσεις από το Ουσμπεκιστάν. Προτού υπάρξει η διεύρυνση της συμφωνίας. Και τα τελευταία χρόνια πολλά βελτιώθηκαν στο Ουσμπεκιστάν, παρότι βέβαια δεν επαρκούν όλα αυτά. Εγώ συγκράτησα από την έκθεση που μας δόθηκε ότι το θέμα αυτό σε σχέση με τα εργασιακά παραμένει ανοιχτό σε σχέση με την forced labor, την υποχρεωτική καταναγκαστική εργασία για παράδειγμα. Και αναφέρεται βέβαια ότι ακόμα και αυτό αν επιτευχθεί δεν επαρκεί και πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω κίνητρα και να βοηθήσουμε να συνδράμουμε το Ουσμπεκιστάν και να συνεισφέρουμε έτσι την κατάσταση στο Ουσμπεκιστάν να την βελτιώσουμε. Είναι όμως πολύ σαφές ότι αν υπάρξουν κάποιες οπισθοδρομήσεις τότε θα έπρεπε να επαναθεωρήσουμε, να ξαναεξετάσουμε αυτή τη στάση μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε όμως το Σμπεκιστάν και την κυβέρνησή του ώστε να μπορέσει να προσχωρήσει σε, ε, να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με τον ΠΟΕ. Και με το πρωτόκολλο αυτό δεδομένων των πολιτικών αλλαγών αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε. Ευχαριστώ για να βοηθήσουμε τους Ουσμπέκους. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατανοώ, οι συντηρητικοί σε αυτή τη φάση δεν θα παρέμβουν. Ο κύριος Πακούλα παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή παρουσίαση. Σε αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια νέα δημοκρατία έχουμε μπροστά μας με το Ουσμπεκιστάν και εμείς ως ε, Ευρωπαίοι θέλουμε τις δημοκρατικές εξελίξεις να τις υποστηρίξουμε και ελπίζουμε ότι οι αρχές και αξίες που είναι σημαντικές για τους Ευρωπαίους, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης οι ελευθερίες, οι πολιτικές θα μπορέσουν να βελτιωθούν στο Σμπεκιστάν και σε σχέση και με τα εργασιακά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο τμήμα. Όταν θέλουμε να προωθήσουμε τα θέματα εμπορίου και διμερώς θέλουμε να διευρύνουμε συμφωνίες με το Σμπεκιστάν. Καλό ήταν το ότι ακούσαμε ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη που ανιχνεύεται στο Ουσμπεκιστάν σε σχέση με την παιδική εργασία για παράδειγμα. Καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η θετική επίπτωση και ότι η δημοκρατία κινείται προς την ορθή κατεύθυνση σε αυτή τη χώρα. Και σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό να δούμε και να εστιαστούμε με αφορμή άλλα θέματα τις προσπάθειές μας να τις εστιάσουμε υπογραμμίζοντας τις δικές μας αξίες ε, στην εμπορική πολιτική αλλά να μην υπάρχουν διπλοί γνώμονες και διπλά σταθμά και μέτρα ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους εταίρους. Μια θετική εξέλιξη λοιπόν ανοιχνεύεται και παρουσιάζεται σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Καλό είναι να συνεχιστεί αυτή. Αναμένουμε στις συζητήσεις με το Ουσμπεκιστάν αυτό να προχωρήσει. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών πρόσφατα ε, είχαμε προβληματιστεί σε σχέση με το θέμα αυτό και ίσως σήμερα σε σχέση με την κυβερνητική αλλαγή θα μπορούσαμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Από το Google δεν γνωρίζω αν ο Ισλάμ Καρίμοφ εξακολουθεί να ε, είναι ε, εν ζωή ή όχι, αν έχει αποβιώσει. Υπάρχουν κάποιες φήμες για κάποιον λέει που θα τον διαδεχόταν. Ε, θα πρέπει να αποσαφινιστούν αυτά και να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της δημοκρατίας ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much and, uh, I... Ευχαριστώ πολύ. Ήγκουε τώρα. Παρακαλώ κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Κόλαφ για την ε, παρουσίασή του που ήταν πλήρης όσον αφορά και την παιδική εργασία και την κατανακαστική εργασία. Ένα θέμα που ήταν κλειδί έτσι κι αλλιώς για το κείμενο που ετοιμάσαμε το 2011 και τις συστάσεις μας. Η κοινωνία των πολιτών και τα αυτόνομα συνδικάτα είναι στοιχείο κλειδί και λένε ότι υπάρχει βελτίωση όσον αφορά αυτά τα θέματα. Είναι μια προπόθεση η κατάργηση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας έτσι κι αλλιώς για το gsp σύν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ποια είναι τα συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις που έχει κάνει ο ΔΟΕ. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, αλλά και άλλοι όπως είναι το Human Rights Watch και άλλοι διεθνείς οργανισμοί ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θέλω να τονίσω πάντως ότι το βασικό για αυτά είναι η βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Μας τα είπε και ο εισηγητής από τον ΔΕ είναι κάτι που μας είπε ότι έχει επιτευχθεί, η βελτίωση αυτή δηλαδή, αλλά πρέπει να εποπτεύουμε κάθε τόσο, να διαπιστώνουμε κατά πόσο ισχύουν και στην κυβερνητική δομή και πιστοποιείται και από τα συνδικάτα. Όλο το σύστημα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία ε, των τομέων του κυβερνητικού, των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών δηλαδή. Η συνεργασία είναι πράγματι αναγκαία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η αυτονομία των συνδικάτων, να προωθωθεί αυτή, να υπάρχει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, στην απεργία. Όλα αυτά πρέπει να είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε τον στόχο που είναι η κατάργηση όχι μόνο της παιδικής εργασίας, αλλά οποιοδήποτε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης, καταναγκαστική εργασία κτλ. Τα εργασιακά δικαιώματα, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν ε, γίνονται σεβαστά, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να καταγγέλλεται αυτό από τα συνδικάτα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει αυτονομία. Το 2016 πάντως ξέρουμε ότι ακόμα πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να ζητήσουν, υποχρεωθούν, υποχρεώθηκαν βασικά να ζητήσουν να δουλέψουν την συγκομιδή αυτή, ε, τελικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν σε εθελοντική βάση πράγματι. Τα εργασιακά δικαιώματα λοιπόν πρέπει να προωθηθούν στη χώρα αυτή με συγκεκριμένες δομές. να υπάρχει ελευθερία του συνεταιρίζεστε και η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα η διεθνή συνεργασία, πρέπει να συμμεριστεί την ευθύνη. Και είναι και δικιά μας υποχρέωση να κοιτάμε τι συμβαίνει και πίσω από τη σκηνή και ποια είναι η δυνατότητα των συνδικάτων όντως να μιλήσουν και να δράσουν. Γιατί πιθανόν το ειδικό καθεστώς μπορεί να τους εμποδίζει να συμμετέχουν σε συλλογικές συμβάσεις. Μέχρι τώρα πρέπει να έχει μια ειδική άδεια κάποιος αν θέλει να ζητήσει μια διαφορετική δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε τι προϋποθέσεις απαιτούνται για να μπορούν οι εργαζόμενοι να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Οποιαδήποτε συμφωνία συνεργασίας λοιπόν πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη αυτά και η Μαρία αρένα πρέπει να καλύψει και αυτά τα κενά που περιέγραψα. Πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο το θέμα της εργασίας, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, Χέλμουτ. Συνεχίζουμε με το EFTD, με τους πράσινους, όχι, ENF, όχι. Ωραία, έχουμε δύο συναδέλφους από την Επιτροπή ΑΦΕΤ που και εκείνη εξετάζει αυτό το θέμα. Συντάκτης γνωμοδότησης, η κυρία Λούνατσεκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Γεια σας, καλή σας μέρα. Και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Ουσμπεκιστάν για την πρόοδο που επετεύχθη από το 2011. Το θυμάμαι, είχα πάει εκεί και υπήρχαν συζητήσεις, οι ανησυχίες ήταν ευρύτερες στο κοινοβούλιο και όταν ψηφίσαμε τότε σε σχέση με 603 ε, μέλη στην Ολομέλεια που υπερψήφισαν και μόνο 8 ήταν εναντίον. Η ανησυχία λοιπόν ήταν τεράστια από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Και σε σχέση με την εκρίζωση της παιδικής εργασίας για τα όσα έχουν γίνει, αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις πράγμα το οποίο κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό πλέον σε σχέση με κάποια χρόνια πριν. Είναι μια πρόοδος αυτή σίγουρα, παρόλα αυτά για την καταναγκαστική εργασία και που αυτό συμπεριλαμβανόταν στο ψήφισμα τότε, η πρόοδος που βλέπουμε και από τα όσα ακούμε από την Άιλο, μάλιστα επετεύχθη πρόοδος σε σχέση με την καταναγκαστική εργασία, αλλά με τα όσα μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης και από διάφορες οργανώσεις και φορείς, είναι ότι ακόμα και σήμερα προετοιμάζει καταλόγους απασχολούμενων δημόσιων οργανισμών για να εργάζονται σε σχέση με το μάζεμα του βαμβακιού και ακόμα και όταν λένε ότι δεν είναι καταναγκαστική συμμετοχή τους, ε, δεν εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν, παρόλα αυτά υπάρχει πρόβλημα αυτό. Και στη Φεργάνα, στην κοιλάδα της Φεργάνα για παράδειγμα, που οδηγούνται ακριβώς εκεί στο, στην κοιλάδα για να μαζέψουν το βαμβάκι. Υπάρχει εκεί ζήτημα. Υπάρχει βέβαια πρόοδος, εντάξει, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω από την ΆΙΛΟ, το Διεθνές Γραφείο, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, να αναμείνουμε μέχρι ότου η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας θα έχει κατατεθεί και θα έχει ολοκληρωθεί. Και μόνο το Δεκέμβριο θα γίνει κάτι τέτοιο, με όλα τα πλήρη στοιχεία και τεκμήρια. Να αναμείνουμε λοιπόν, διότι νομίζω τότε θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει και βρίσκεται υπό εξέλιξη. Συμφωνώ, υπάρχει πρόοδος και είναι αυτό κάτι που μας ικανοποιεί. Εντάξει, όμως παρόλα αυτά από τα όσα έχουμε ως στοιχεία που μας διαβιβάζονται δεν νομίζω ότι αυτό επαρκεί. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε πει στην έκθεσή μας του 2011 είχαμε πει κάθετα και το αναφέρω ως παράθεμα ότι θα πρέπει εδώ σημαντικά αποτελέσματα να επιτευχθούν ώστε να ξεριζωθούν η καταναγκαστική εργασία και η παιδική εργασία, να εξαλειφθούν. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα ζήτημα, κάποιο κενό. Θα ήθελα να προτείνω και γνωρίζω ότι οι συντονίστες αποφάσισαν ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την ψήφιση ε, και για το Δεκέμβριο. Θα ήθελα να σας ζητήσω, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ξεκινάει τώρα η συζήτηση για αυτά τα θέματα, θα ήθελα να το αναβάλουμε για ένα μήνα, ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να λάβουμε άλλα στοιχεία και τα θέματα αυτής της έκθεσης. Ένας μήνας δεν είναι τεράστιο πρόβλημα, νομίζω. Ελπίζω τουλάχιστον, ευελπιστώ ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και θα ήθελα να πω, δεν πρέπει να βιαζόμαστε ή να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ένας μήνας πάνω κάτω δεν κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Διότι παρότι συμφωνώ τα μάλα ότι το Κοινοβούλιο ειδικά Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρόεδρος, τι συμβαίνει ακριβώς και με την πολιτική κατάσταση εκεί που βρίσκεται εν ρευστό. Λοιπόν, 25 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της χώρας αυτής σημαντική, σημαντικό ορόσημο αυτό για τους πολίτες του Μπεκιστάν ούτως ή άλλως παρόλα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε πώς να το τις θέσεις μας ώστε να επιτηρήσουμε, να επαγρυπνούμε για ε, το τι συμβαίνει και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκ του σύνεγγης. Και κάποιες ερωτήσεις άμεσα προς, προς τον Άιλο. Είπατε, αναφέρατε ότι ναι, μια μεγάλη πλειοψηφία πολιτών εθελούσια καταλήγουν στη συγκομιδή αυτή. Σε μια κατάσταση όμως, σε μια χώρα όπου υπάρχει μεγάλη καταστολή, μεγάλη καταπίεση, πώς μεθοδολογικά μπορείτε να το πείτε αυτό ότι μπορεί να διασφαλιστεί ότι με καταθέσεις ατόμων που λένε ότι εθελούσια συμμετέχουν κάτι τέτοιο αποδεικνύεται. Είναι δύσκολο με ένα τέτοιο καθεστώς να πει κανείς αν κάτι τέτοιο συμβαίνει ή όχι. Είναι και θέμα μεθοδολογικό. Πώς ρωτά κανείς κάποιον για να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Είσαστε εσείς μόνοι, μόνοι σας σε αυτές τις συνεντεύξεις ε, και επαφές με αυτές τις καταθέσεις ε, από τους πολίτες του Ουσμπεκιστάν να μπορούν ε, υποκαθεστώς εχεμήθειας να σας εμπιστευτούν κάτι τέτοιο. Και υπό την περιβαλλοντική πτυχή επιπλέον θα έπρεπε εμείς ως Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε κάπως ε, στην πολυμορφοποίηση της γεωργίας, να μην είναι μονοκαλλιέργεια το βαμβάκι στο Ουσμπεκιστάν ή και αλλού, όπως υπάρχει το ζήτημα των μονοκαλλιεργειών και ένα πρόβλημα. Και το θέμα της άρδευσης δημιουργεί πρόβλημα για την ίδρευση των πολιτών, μια και όλο το νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση του βαμβακιού. Με την ανάλυση όλων αυτών των πραγμάτων ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε αναμένοντας να κατατεθούν τα, να είναι διαθέσιμα τα τεκμήρια και από την άλλο και, άλλο και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφος Κούκαν τώρα που είναι σκιώδης εισηγητής και αυτός για το ΕΛΚΑ στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Έχετε τον λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ας ξεκινήσω αναφέροντας ότι από το ΕΛΚΟΣ και όδηση συγητής για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Η εμπλοκή σε σχέση με τις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κέρια σημασία πιστεύω ότι θα έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερα στις προσπάθειές μας για τις χώρες αυτές από πλευράς του Κοινοβουλίου. Μια και κάθε χώρα είναι διαφορετική και έχει τις δικές της ιδιομορφίες, χρειάζεται εξειδικευμένη προσέγγιση για κάθε χώρα αυτής της περιοχής. Και για αυτό το χαρτοφυλάκιο πρώτον Είμαι πεισμένος ότι περαιτέρω εμπλοκή και συμμετοχή με την κυβέρνηση και τις αρχές του Ουσμπεκιστάν είναι θεμελιώδους σημασίας. Αναγνωρίζοντας τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί, μπορεί κανείς να συμφωνεί, ή να διαφωνεί, παρόλα αυτά όμως είτε είναι μεγάλη πρόοδος, είτε μικρή, είτε περιορισμένη. Πρόοδος όμως διαπιστώνεται ότι υπάρχει. Και νομίζω ότι κατά τον έναν ή άλλο τρόπο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη χώρα να προχωρήσει και εξετάζοντας εκ του σύνεγγυς πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Με τέτοιο τρόπο ώστε να γνωρίζουν οι Ουσμπέκοι ότι εμείς ε, βρισκόμαστε πραγματικά σε γρήγορση. Τώρα, σε σχέση με την έκθεση όσον αφορά το 2015, από το φθινόπωρο του 2015, θα πρέπει να ε, είμαστε πιστοί στην ε, υπόσχεσή μας να ξανανοίξει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Πρέπει να έχουμε μια συμβατική σχέση με τη χώρα αυτή όσον αφορά τα κλωστοϊφαντουργικά επίσης. Και όσον αφορά αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Τώρα για την αναβολή της ψήφισης χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί. Τα τελευταία τρία χρόνια υπήρχε μια στρατηγική όλων αναβολών, αναβολών και νέων αναβολών. Να είναι αυτό η σωστή πορεία δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη στρατηγική. Βρισκόμαστε σε αρχές Σεπτεμβρίου 2016. Να λέμε τώρα να αναβάλουμε για ένα μήνα, κατανοώ Ρίκε... Λούνατσεκ τους πρακτικούς λόγους για τους οποίους αναφέρει σε αυτό το επιχείρημα. Αλλά αν φτάσουμε και όταν φτάσουμε το Δεκέμβριο μήπως υπάρξουν και άλλοι λόγοι για παράδειγμα πρόεδρος, κυβέρνηση κτλ. Και πάλι αναβάλουμε και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ΕΣΑΗ στο Δινεκές. Θα πρέπει να υπομισθούμε περισσότερες ευθύνες πιστεύω όχι να λάβουμε τώρα κάποια απόφαση να αναβάλουμε, να τηρήσουμε την αρχική ε, προθεσμία του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλος να ζητά τον λόγο από τα, τους ευρωβουλευτές για να εκφράσει τις απόψεις του. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς που είσαστε επικεφαλής της ε, μονάδας στην Γενική Διεύθυνση, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να υπενθυμίσω σύντομα το πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής για τις σχέσεις μας με το Ουσμπεκιστάν δηλαδή, όπου υπάρχει μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασίας από το 1999 και το ο κείμενο ήταν εκτός ε, του GSP. Ήταν μια διμερής συμφωνία μέχρι το 2004. Από το 2004 που εξέπνευσε η συμφωνία αυτή δεν υπήρξε κάτι άλλο για την υφαντουργία. Το πρωτόκολλο σήμερα έχει στόχο ακριβώς να τροποποιήσει την συμφωνία προκειμένου να συμπεριληφθεί και η υφαντουργία στο πεδίο εφαρμογή. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα διευκολυνθεί το εμπόριο και ιδιαίτερα υπέρ νέων εξαγωγών ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε εδώ για έναν τομέα όπου οι εμπορικέ ροές είναι πολύ περιορισμένες όσον αφορά το παπάκι από το Σπίκιστάν, που είναι η έκτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα και η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγέας βαμβακιού αλλά 54 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι εξαγωγές σε μας από το 1 εκατομμύριο συνολικά από το Ουσβεκιστάν. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και πολύ χαίρεται που βλέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Ουσβεκιστάν και τον ε, ΔΟΕ. Εμείς δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια. Ιδίω από το 2011, όταν υιοθέτησε το ψηφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου η συνεργασία αυτή να καταστεί πράγματι εφικτή, πράγμα το οποίο έγινε το 2013. Και εκφράσουμε την ικανοποίησή μας επίσης που βλέπουμε ότι παίρνει μια πιο συγκεκριμένη δομή η συνεργασία αυτή. Μια συνεργασία όπου συμμετέχουν όλο και περισσότεροι και από τις δύο πλευρές. Οι εκπρόσωποι του ΔΟΕ μόλις είπαν ότι υπήρξαν διάφορα προγράμματα στήριξης, ε, την εργασία το 2016, το πρόγραμμα δράσης το 2016 για τα επόμενα χρόνια προκειμένου να καταργηθεί καταναγκαστική εργασία και τώρα και ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες έχουν εκπονηθεί από πλευράς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Και εμείς λοιπόν για το μέλλον υποστηρίζουμε μια τέτοια συνεργασία. Καλωσορίζουμε επίσης και τις θετικές ε, εξελίξεις που έχουμε διαπιστώσει επί τόπου. Όπως είπατε, πολλοί από εσά έχει επιτευχθεί πράγματι σημαντική πρόοδος για να καταργηθεί η παιδική εργασία. Και υπάρχει πρόοδος και στο θέμα της καταναγκαστικής εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας που μας συνόψεις εδώ δείχνουν ότι υπάρχει μια θετική τάση. Εννοείται ότι όλοι είπαμε και λέμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Πέρα δηλαδή από διάφορες δράσεις οι οποίες ήδη έγιναν τη χρονιά που πέρασε. Υπήρξε μια εκστρατεία συνειδητοποίηση του κοινού, υπήρξε επίσης μια διαδικασία προκειμένου να έχουμε την άποψη του κοινού, του κόσμου, της κοινωνίας. Οπότε φτάνω στο τελευταίο μου σημείο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από πλευράς Κομισιόν, εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεχίζεται όσον αφορά το κείμενο του πρωτοκόλου και ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα. Μέσα στο 2016 δηλαδή, αν μη τι άλλο. Και θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε την Επιτροπή σας για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε επαφή με τις αρχές του Ουσμπεκιστάν προκειμένου να επαναλάβει τη σημασία που δίνουμε στην κατάργηση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε δραστήριοι επίσης και με τον ΔΟΕ και να στηρίζουμε τις προσπάθειές του για τον έλεγχο και την εποπτεία της κατάστασης επιτόπου. Επιτρέψτε μου επίσης να σχολιάσω κάποια πράγματα που υπόθηκαν για την διαφοροποίηση της οικονομίας του Ζουβεκιστάν. Είναι κάτι που στηρίζουμε και εμείς και συνεργαζόμαστε με τις αρχές της χώρας έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και για να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες πέρα της γεωργίας. Δουλεύουμε λοιπόν πράγματι πάνω σε όλα αυτά για να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας. Εννοείται. Το μπαμπάκι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μειώνεται κάπως σαν παραγωγή, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η τάση διαφοροποίησης ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τόσο μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μήπως έχει σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχω κάποια σχόλια, γιατί τα περισσότερα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Πρώτον, όπως θα θυμόσαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο διότι φρόντισε ήδη πριν από 3-4 χρόνια να οθήσει προς την κατεύθυνση αυτή της προσέγγισης ανάμεσα στο Διεθνές Οργανισμό Εργασίας και του Σμπεκιστάν. Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα εξαιτία της κατάστασης, αλλά ε, το έργο προχώρησε. Και τώρα ενισχύεται αυτή η συνεργασία, κάτι το οποίο εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος. Στηρίζουμε πάντα πολύ το εξαιρετικό έργο του ΔΟΕ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Αν κοιτάξουμε ευρύτερα την εικόνα, το Σβεκιστάν είναι μία από τις λίγες χώρες όπου έχει επιτεθεί τόσο μεγάλη πρόοδος για ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι η καταναγκαστική και παιδική εργασία και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι που πρέπει να εκτιμήσουμε και να ανταμείψουμε. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η δουλειά μας. Όχι, σίγουρα μένει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα, το είπαμε όλοι. Και θα παραμείνουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί να δούμε τι πρόοδος θα επιτευχθεί φέτος, για παράδειγμα. Έχουμε ακόμα τη δυνατότητα, αν χρειαστεί, να στηρίξουμε τον έλεγχο του ΔΟΕ όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και του χρόνου, αν χρειαστεί. Αν χρειάζεται κάποιος από εσά την ε, καθησύχασή μας ότι δεν σταματάμε αλλά συνεχίζουμε, ε, τον έλεγχο, να ξέρετε ότι γίνεται. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη μας τις τάσεις των τελευταίων τριών ε, τεσσάρων ετών, υπάρχει μια σταθερή θετική τάση. Χωρίς να λέω ότι σταματάμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε αν χρειαστεί τα επόμενα χρόνια. θα συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία. Τώρα, για να πάμε πίσω στο 2011, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε. Αυτά τα οποία διαβάσαμε τότε ήταν ότι το Σουβεκιστάν θα πρέπει να είναι στην διαδικασία κατάργησης της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας λίγο πολύ το πετύχαμε, γιατί η παιδική εργασία έχει περίπου καταργηθεί και η καταναγκαστική εργασία είναι στη διαδικασία κατάργησης. Σημαντικά αυτά. Και δύο τελευταία λόγια. Η συνεργασία με το Σμπεκιστάν περιορίζεται στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν από πλευράς ε, συνεργασίας να βοηθήσουμε και σε αγροτικές μεταρρυθμίσεις και αγροτική διαφοροποίηση, ώστε να μην περιορίζονται στην μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού. Και αυτά σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με την οποία συνεργαζόμαστε επιτόπου. Έτσι, έχουμε κάθε λόγο να ελπίσουμε ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και θα αποφέρει καρπούς συντομότατα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τα σχόλια αυτά και είναι προφανές ότι όντως το πανόλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι οργανισμοί εδώ ότι το βασικότερο είναι η παιδική εργασία και η καταναγκαστική εργασία όπως μας είπε και ο κύριος Κόλλερ, οπότε θα του ξαναδώσω το λόγο για να απαντήσει <coughs> στις ερωτήσεις και σε ό,τι σχόλια έγιναν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για την εκτίμηση του έργου μας όπως εκφράσατε στις παρεμβάσεις σας που ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις πρωτού δώσω τον λόγο στον κύριο Ταμπιόλα που ήταν παρόν εξ αρχής και είναι ο πραγματογνώμων μας επί του θέματος. Θα ήθελα να ξανατονίσω εδώ ότι ξεκινήσαμε το 2013 με τις εργασίες μας εκεί και σε τρία χρόνια όλα και όλα μπόρεσε να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχει αλλάξει και η νοοτροπία, η προσέγγιση από το ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε μια πιο πρόθυμη συνεργασία και τριμερή συνεργασία, πολυμερή συνεργασία και σε σχέση με την ε, επικύρωση θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας ε, στο πρόγραμμα εργασιών μας. Επιτρέψτε μου να εκφραστώ στο ότι θα πρέπει με αυτή την τάση που έχει σημειωθεί να δώσουμε συνέχεια και θα πρέπει να διευρύνουμε και τη συνεργασία μας και να την εντάξουμε σε μια ευρύτερη προσέγγιση για ένα πρόγραμμα για τη χώρα αυτή. Και υπάρχουν και πολύ θετικά μηνύματα σε σχέση με αυτό από τους εταίρους μας στο Ουσμπεκιστάν. Όσον αφορά τη δημοσίευση της έκθεσής μας, ο Δεκέμβριος θα ήταν ίσως και η πιο πρώιμη ημερομηνία για να επιτευχθεί αυτό. Πρέπει φυσικά να συνεργαστούμε και με τους εταίρους μας στο Ουσμπεκιστάν για να ολοκληρώσουμε. Είναι, ας το πω έτσι, μια πολύ αισιόδοξη πρόπτικη να δημοσιευθεί το Δεκέμβριο, αλλά θα προσπαθήσουμε, αν γίνεται, να το πετύχουμε αυτό. Ο κύριος Ταπιόλα τώρα θα έχει τον λόγο για τα άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς σε όλη αυτή την εποπτική διαδικασία ότι έχουμε καταλήξει σε μια νέα φάση πλέον. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής προοπτική μέσα σε αυτή τη συμφωνία για το πώς διαμορφώνεται και πώς έχει η κατάσταση. Η αρχική εποπτεία και επιτήρηση αφορούσε τη διαπίστωση του πώς ακριβώς είχε η κατάσταση επιτόπου γιατί υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ε, επί του θέματος. Τώρα, έχοντας ε, κοιτάξει, έχοντας προσέξει τι συμβαίνει ακριβώς και έχοντας και μια ποσοτική ε, δειγματοληψία πέρα από την επιτήρηση ως διαδικασία μπορούμε τώρα να επικεντρωθούμε στο να καταλήξουμε στο να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια για την εξάλληψη της παιδικής εργασίας διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιστρέψει το φαινόμενο της παιδικής εργασίας από ε, την πίσω πόρτα και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους ε, της ε, καταναγκαστικής εργασίας ως φαινομένου στο Ουσμπεκιστάν αναφέρθηκε. Μία από τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν αφορούσε τις παρατηρήσεις του Human Rights Watch. Είχαμε συζητήσεις σε σχέση με την οργάνωση αυτή Human Rights Watch και σε σχέση με τη συγκομιδή του Βαμβακιού. Υπήρξαν εξηγήσεις ε, και δεν νομίζω ότι έχουμε και πολύ διαφορετικές απόψεις επ' αυτού για το πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Εμείς όπως ε, ανέφερε ο κύριος Κόραρ έχουμε πολλούς ε, που εθελοντικά δηλώνουν εθελούσια ότι καταλήγουν στη συγκομιδή βαμβακιού. Υπάρχει και μία, ας το πω έτσι, λόγω της κοινωνικής πίεσης, ε, μία μικρότερη προθυμία ίσως υπάρχει μια διαδικασία την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε σίγουρα επικεντρωνόμενοι σε αυτά με τους εταίρους μας τους Ουσμπέκους είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει επίκεντρο εστίασης της επιτήρησής μας, της εποπτείας μας. Μέσω της εποπτείας επιτήρησής μας εξετάζουμε πώς οι πρακτικές αυτές μπορούν να τροποποιηθούν, να μεταβληθούν. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους μεταβολές και πώς θα μπορούσαν οι διάφορες οι διαφορετικές εκστρατείες και τα μηνύματα που διαχέονται και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα μπορούσαν να τελεσφορήσουν. Είναι κάτι επί το οποίο συνεργαζόμαστε με τους Ουσμπέκους εταίρους μας, ομολόγους μας και φυσικά και με συνεργαζόμαστε και του σύνεγγις και με την εποπτεία αυτή σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα. Ε, αυτό με οδηγεί και στο θέμα του συγχρονισμού, του, της χρονικής πτυχής των θεμάτων για την συγκομιδή που ε, κατά τον Οκτώβριο ή τέλειο Οκτωβρίου τέλος πάντων θα έχουμε τη δυνατότητα, θα θέλαμε να ε, συντάξουμε μια έκθεση το Νοέμβριο, κατά τέλη Νοεμβρίου και στην Παγκόσμια Τράπεζα και στην ομάδα επαϊόντων του ILO. Θα είναι μια χρονική στιγμή αυτός ο συγχρονισμός που θα μπορούσαμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα για το πρόσφατο παρελθόν, για το τι έχει σημειωθεί και επισυμβεί εκεί. Η διαδικασία είναι σίγουρα κάτι το οποίο ούτως ή άλλως παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης για παράδειγμα σε σχέση με τα δειγματοληπτικά στοιχεία που έχουμε και που αποτελούν τμήμα της ε, συνολικής διαδικασίας αποτελούν τμήμα της ευρύτερης αυτής προσέγγισης σε σύγκριση με το 2014-2015 βασίζονται όλα αυτά σε σχέση με τα στοιχεία που μας δίνονται από συνεντεύξεις βέβαια συνεργαζόμαστε με ουσμπέκους εταίρους όχι τους κυβερνητικούς εταίρους αλλά με την τους ε, επαΐοντες και οι δήμονες ε, της ε, ουσμπεκικής πλευράς. Όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία αναλύονται και σταθμίζονται βρίσκονται στα χέρια του ILO. Φυσικά γίνονται και συνεντεύξεις σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα ή ζητήματα ως ερωτήματα και οι απαντήσεις που μας παρέχονται και αυτές αναλύονται. Πρέπει να, να δούμε αν υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν έτυχαν απαντήσεων, θέματα τα οποία δεν απαντήθηκαν επαρκώς, αλλά η αναλογία σε σχέση με εκείνους που απάντησαν είναι πολύ υψηλή ο, βαθμός εκείνων που, ο αριθμός εκείνων που απάντησαν είναι πολύ υψηλός με την ανάλυση και την επεξήγηση που θα γίνει θα έχετε την ευκαιρία του χρόνου, νωρίς του χρόνου 2017, να έχετε αυτά τα στοιχεία στα χέρια σας. Okay, thank Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και... Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για τη συνεργασία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και με τα, ε, τις διεθνείς οργανισμούς. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση σας δίνοντας το λόγο στην εισηγήτρια. Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αρκετά πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούσαμε όσον αφορά το περιεχόμενο. Πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί, ε, διαφορετικά επίπεδα. Ακούσαμε ομόφωνα αναγνώριση για τις προσπάθειες που έγιναν όσον αφορά την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία, σε διαφορετικά επίπεδα βεβαίως. Ε, κάποιοι αναγνωρίζουν ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος, κάποιοι άλλοι έχουν και κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το επίπεδο της πρόοδου, αλλά γενικότερα όλοι θεωρούν ότι υπήρξε πρόοδος. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι επίση σημαντικό να διαβάσουμε το μήνυμα ότι Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται διαμιάς. Είναι μια συνεχής διαδικασία ώστε το Ουσμπεκιστάν να συνεχίσει ε, και σε θέματα προστασίας παιδιών αλλά και σε θέματα προστασίας εργαζομένων. Θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό και το είπα και προηγουμένως να μπορούμε αφενός ε, να ε, επικροτούμε τις, ε, τα θετικά στοιχεία, αλλά και να σταθούμε και στα αρνητικά μέσω ενός ψηφίσματος, διότι η παράταση ενός πρωτοκόλλου κλωστοφαντουργίας δεν μας επιτρέπει να εκφράσουμε όλες μας τις επιφυλάξεις. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψήφισμα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και τα επιχειρήματά μας, αλλά και να αποστείλουμε και ένα πολιτικό μήνυμα ε, προς τις Ουσμπεκικέ αρχές για να μπορέσουμε και να προσδώσουμε αξία στα όσα έχουν κάνει μέχρι τούδε, αλλά και για να του ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσουμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα, να απαντήσουμε δηλαδή το συντομότερο δυνατόν για αυτό το πρωτόκολλο για την κλωστοφαντουργία, θα ήθελα να ζητήσω να μπορέσουμε να έχουμε και μία απόφαση στους συντονιστές ε, της Επιτροπής μας ε, για το ψήφισμα. Ε, θα καθορίσει και τι πρέπει να κάνω εγώ ως εισηγήτρια και φυσικά να μπορέσουμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εκφράσουμε και ε, όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Κανείς δεν είπε ότι όλα είναι τέλεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αποστείλουμε και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ε, ενώπιον των ουσμπεκικών αρχών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ψήφισμα, επομένως χρειάζομαι και την απόφαση αυτή. Ευχαριστώ. Βεβαίως δεν είναι δική μου δουλειά εδώ να έχω άποψη ως προς το χρονοδιάγραμμα. Οι συντονιστές θα αποφασίσουν και θα πρέπει λοιπόν να παραπέμψω το θέμα αυτό στους συντονιστές. Προς το παρόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στο παρόν είναι ότι 12 και 13 Οκτωβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, αλλά ε, θα το παραπέμψουμε το θέμα στους συντονιστές και θα αποφασίσουν στην επόμενη συνεδρίασή τους. Με αυτό ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 22, σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών. είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για το θεματολόγιο της ε, Επιτροπής μας. Έχουμε και μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, ε, την οποία έχει αναλάβει η συνάδελφος η Έμα Μακλάρκιν και η οποία είναι συντάκτηρα και της γνωμοδότησης. Να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και ελπίζω να έχουμε και σκιώδεις συζητητές, ε, το πρόγραμμα δράσης για την προστασία των άγριων ειδών είναι ένα πρόγραμμα... Ο Πρόεδρος Διακόπτη, σα παρακαλώ λίγο ησυχία για να ακούσουμε την εισηγήτρια. Ό,τι συζητήσεις έχετε, παρακαλώ εκτός αιθούση. Ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρο. Έλεγα λοιπόν ότι το πρόγραμμα προστασίας άγριων είναι μια πολυδιάστατη προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα κατά των άγριων ζώων. Παράνομο εμπόριο βεβαίω αυτών των αγαθών και αυτό το πρόγραμμα δράσης αναγνωρίζει τη σημασία συνεργασίας ε, και ευθυγράμμισης των ε, προτεραιοτήτων του εμπορίου για να καλύψουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και τι σχέση υπάρχει με τη γνωμοδότηση αυτή προς την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη δική μας έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο, που θα πάει πολύ πιο πέρα και θα σταθεί σε τεχνικά θέματα εμπορίου στο θέμα αυτό. Έχουμε μία ε, άνευ προηγουμένου αύξηση εμπορίου παρα, ε, νόμου αγρίων ειδών και το εμπόριο αυτό και οι εγκληματικές δραστηριότητε οδηγούν σε 8 ε, με 20 δισεκατομμύρια ευρώ ε, Ετησίω και από την ε, απογραφή που έγινε για τους ελέφαντε διαπιστώνεται ότι υπήρξε τεράστια απώλεια στην Αφρική ελεφάντων. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιε συνέπειε, όχι μόνο προ τη βιοποικιλότητα αλλά υπάρχουν και πολύ άσχημε συνέπειε όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση σε ε, ξένες χώρε. Ε, συνδυάζοντας αυτό λοιπόν με την αποσταθεροποίηση της ασφάλειας σε διάφορες χώρες, δεν μας ενδιαφέρει απλώς η περιβολατική προστασία, αλλά μας ενδιαφέρει ε, και το γεγονός ότι χάνεται μια πηγή χρηματοδότησης για το οργανωμένο έγκλημα. Κατά την εξέταση της γνωμοδότησης θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να σταθούν κυρίως στο πρόγραμμα δράσης και τα υπόλοιπα στοιχεία να τα κρατήσουμε για την έκθεση της Επιτροπής μας που θα σταθεί σε μηχανισμούς εμπορίου που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε μέτρα ως τμήμα των πολιτικών εμπορίου και των συμφωνιών για να τηρήσουμε τους στόχους βιωσιμότητας. Η έκθεση του Δεκεμβρίου θα προβάλλει διεθνείς συνθήκες και οργανώσεις όπως για παράδειγμα το BOE, τις σάιτες, ε, το OECD και το UNEP. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε τμήμα ενός διεθνούς καθοριστικού κινήματος και να φροντίσουμε να έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές που χρειαζόμαστε διακαώς. Επίσης θα εξετάσουμε ε, την πολιτική και θα δούμε και την αξιολόγηση της παρούσας εφαρμογής των κεφαλαίων της βιώσιμης ανάπτυξης στην κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση, εδώ θέλουμε να έχουμε δεσμού μεταξύ αρκετών κλάδων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια διπυρωτική απάντηση στο, ε, σε αυτή τη μορφή εγκλήματο. Το σχέδιο γνωμοδότησή μου, λοιπόν, επικεντρώθηκε σε τέσσερι τομεί. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό από πλευρά ε, ε, Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου να ενθαρρύνουμε την καλύτερη χρήση των ε, πόρων που έχουμε στη διάθεσή μα αυτή τη στιγμή. Όπω για παράδειγμα παρακολούθηση, κατάρτιση για τελωνιακέ αρχέ σε χώρε προορισμού και διέλευση και φυσικά να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν αυτή τη μορφή εμπορίου. Δεύτερον, θέλουμε κάποιε διατάξει για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ε, για να υπάρχουν σε οποιοδήποτε σχέδιο, όχι μόνο σε εμπορικέ συμφωνίε, αλλά και κατά την. Ε, οποιαδήποτε αναπτυξιακή βοήθεια δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτόν τον αγώνα. Ε, υπάρχουν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, δίκτυα διανομής, ε, οργανώσεις μεταφορέων και ε, επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, επομένως πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση. Και τέλος πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συμβατότητα με τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίου του ΠΟΕ. Το πρόγραμμα ε, άγριας ε, ζωής ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα σε σχέση με διεθνεί συμφωνίες ή διεθνείς εκστρατείες για την καταπολέμηση αυτή τη μορφή εμπορίου. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε αυτό το πεδίο εφαρμογή και ίσω θα μπορούσατε να καταθέσετε τροπολογίε που μα ενδιαφέρουν περισσότερο να μην ξεπεράσουμε τα όρια εδώ, να σταθούμε στα όρια και να δούμε την έκθεση η οποία θα υποβληθεί αργότερα, η οποία θα έχει τα υπόλοιπα στοιχεία. Ε, θέλω λοιπόν να ε, δεσμευθούμε για το πρόγραμμα ε, για την άγρια ζωή του Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή τη γνωμοδότηση αλλά και στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ο κύριος Βάνσον και όδες εισηγητές πρώτα το Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους του κύριου Φιέλνερ που είναι σκιώδης εισηγητής έχω να σας διαβάσω ταξίς. Πολύ καλή γνωμοδότηση της συγγήτριας, της συντάκτρια και πολύ καλή και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε που επικεντρώνεται στα βασικά όσον αφορά την προστασία ε, από το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υπάρχει η συμφωνία από πλευρά του ΠΟΕ και είναι καλό να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι να εμποδίσουμε το παράνομο εμπόριο, αλλά να διευκολύνουμε το νόμιμο εμπόριο. Και για να γίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τρόποι, μεταξύ άλλων να είναι λιγότερο κερδοσκοπικό το παράνομο εμπόριο, που σημαίνει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά, όπως λέει και η συντάκτρια. Η προστασία της άγριας ζωής είναι κάτι πολύ σημαντικό για πάρα πολλές χώρες και δεν θα πρέπει σε αυτές μόνο να βάλουμε το βάρος της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Ευχαριστούμε, David Μάρτιν, τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όπως είπε και Έμα, εδώ δεν πρόκειται μόνο για την προστασία της άγριας φύσης, πρόκειται για την προστασία των φυσικών πόρων στην Αφρική κυρίως. Διότι καταλήγει τελικά η όλη υπόθεση και σε λαθρεμπόριο διαμαδιών κλπ. Το λαθρεμπόριο έχει αυξηθεί μετά τη συμφωνία ΣΥΤΕΣ Έχουν ε, γίνει πολλά. Έχει επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαβάσαμε ένα άρθρο σήμερα το πρωί στις εφημερίδες, που λέει ότι έχουν χάσει τα Ζανία και άλλες χώρες 5% των ελεφάντων τους και στο Κονγκό επίσης. Πολύ σοβαρή κατάσταση. Εγώ συμφωνώ με τα κύρια που λέει η Έμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εκθέση αυτή. Δεδομένου ότι διαπραγματευόμαστε διάφορες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, να αναφερθούν οι χώρες ΑΣΕΑΝ στη γνωμοδότηση και να πούμε ότι σε αυτές τις συμφωνίες με τις χώρες ΑΣΕΑΝ πρέπει να υπάρχουν διατάξεις για την προστασία της άγριας ζωής. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς είναι μία από τις κύριες αγοράς, αγορές τέτοιων παράνομων προϊόντων ε, άγριας ζωής. Γι' αυτό θα πρέπει και εδώ να κάνουμε περισσότερα πράγματα με πιο αυστηρούς ελέγχους στα τελωνία για να καταπολεμήσουμε και εμείς το λαθρεμπόριο αυτό. Και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και ο ΠΟΕ έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο να διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε στη συνεργασία μεταξύ ΠΟΕΣ, ΣΥΤΕΣ, προσφέρουμε τεχνική βοήθεια, να βοηθήσουμε στην ενίσχυση ικανοτήτων κλπ. Η επόμενη συνάντηση ΣΥΤΕΣ θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου στο Γιωχάννεσμπουργκ. Και εκεί θα συζητηθεί πρόταση για να συμπεριληφθεί όλος ο πληθυσμός Άγριας Πανίδας στο παράρτημα 1. Άρα και το ελεφαντοστού θα συμπεριληφθεί και σημαίνει ότι θα απαγορευτεί κάθε τέτοιο εμπόριο. Άκουσα, ελπίζω να μην αλήθεια, ότι ήταν κατά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί αλλά ελπίζω να πούνε ότι θα στηρίξουν την αλλαγή αυτή. Τέλος, μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό είναι ότι η Γαλλία θέλει να απαγορεύσει το εμπόριο και ελεφαντοστού αλλά και από ρινόκερους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, υπάρχει πρόταση να γίνει απαγόρευση αυτή η ευρωπαϊκή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλντε Τακούλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα δράσης αυτό και μια αξιολογή ε, γνωμοδότηση από πλευράς της ΕΜΑΣ. Από ό,τι φαίνεται αυτά τα θέματα, αυτά τα ζητήματα ευρύτερα θα πρέπει τώρα να τύχουν συζήτησης Φυσικά η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε με ιδιαίτερο τρόπο. Η ε, κατάσταση σε σχέση με τα ζώα δείχνει ότι υπάρχει μια μεταβολή και εδώ πολλά πράγματα αναφέρονται σε σχέση με το νόμιμο εμπόριο και σε σχέση και με την ηθική διάσταση του εμπορίου αυτών των ε, προϊόντων. Η σημερινή συζήτηση η οποία διεξάγεται για ένα νέο πρόγραμμα δράσης, ε, όχι μόνο ένα νέο πρόγραμμα δράσης, αλλά την καταπολέμηση ως πρωτοβουλία, καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, ε, εντάσσει πολλά ζητήματα μέσα στο πλαίσιο αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πολύ συχνά διεξάγεται μέσω τέτοιου είδους δραστηριοτήτων και κατά τα τελευταία έτη πρόσφατα μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε αυτό και γι' αυτό θα επιθυμούσα αυτό το πρόγραμμα δράσης να είναι ένα μέσο καταπολέμησης της τρομοκρατίας ακριβώς και κυρίως καταπολέμησης της, ε, ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με αυτό το πρόγραμμα δράσης πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν υποχρεώσεις από ε, να καταργήσουν, να εξαλείψουν αυτό το παράνομο εμπόριο και να καταπολεμήσουν την ε, ανομία και τα, την, τις εγκληματικές δράσεις και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Η γνωμοδότηση από πλευράς της έμας ε, ήταν η πολύ ισορροπημένη και πιστεύω ότι θα έχουμε και μια πολύ θετική έκθεση στην οποία θα καταλήξουμε. Έχουμε Βρετανούς εισηγητές και αυτό είναι ένα ε, χαρακτηριστικό στοιχείο. Ε, θα πρέπει να ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια των επομένων ετών αυτό θα εξυπηρετήσει την Ένωση. Ευχαριστώ. Uh, Σα ευχαριστούμε και τώρα εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μακλάρκιν για την πρότασή της. Ε, συμφωνώ με κάποιες από τις προτάσεις της και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάνε για τον αυτοματισμό χρηματοδότησης. Πρέπει να δούμε όντως πώς θα χρηματοδοτήσουμε εμείς όμως την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Επίσης, πράγματι πρέπει να έχουμε επίκαιρα στοιχεία, ενημερωμένα και χρειάζεται τα τελωνία να ενισχυθούν για την καταπολόμηση της διαφθοράς. Δυσκολεύομαι όμως κάπως να συμφωνήσω με αυτά που λέει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η προστασία από αυτό το παράνομο εμπόριο. Ευχαριστώ. Με συμφωνίες δηλαδή που λέει εμπορικές. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κυρία Μανουέλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την Επιτροπή σας και κυρίως την εισηγήτριά σας που δίνετε τόσο σημασία στο θέμα του παράνομου εμπορίου ε, ειδών που κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Η κατάσταση είναι πράγματι ανησυχητική. Αυτό το υπενθύμησαν πολλοί ευρωβουλευτές σήμερα. Ακόμα και προχτές ε, οι συνάδελφοι από τις κάτω χώρες κατάσχεσαν δύο τόνους προϊόντων που προέρχονται από είδη ε, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Και όλα αυτά με 500 εκατομμύρια ευρώ συνοδευόντουσαν. Όλα αυτά δείχνουν την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο αυτό. Το Συμβούλιο έχει εξετάσει αυτό το θέμα και έχει δώσει τη στήριξή του από τον Ιούνιο που μας πέρασε. Η συνεργασία είναι πράγματι ζωτική σημασίας σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και με την Europol, την Eurojust γιατί πρέπει συλλογικά να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε αυτό το φαινόμενο. Η διεθνή συνεργασία και τα εμπορικά ζητήματα και αυτά έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό υπενθυμήθηκε. Υπήρξε διάσκεψη των μερών της ΣΥΤΕΣ, Μέλλον θα υπάρξει, αυτή που θα γίνει στην Νότια Αφρική, πολύ σύντομα, και αυτή θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία ώστε οι 183 χώρες να συμφωνήσουν για το πώς θα καταπολεμήσουν αυτή τη μάστιγα. Και τη διαφθορά βέβαια. Ρωτήσατε για το ελεφαντοστού, για τους αφρικανικούς ελέφαντες. Επ' αυτού έχω να σας απαντήσω το εξή. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ΣΥΤΕΣ θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν δηλαδή οι συζητήσεις γίνονται, θα υπάρξει και προφορική ερώτηση σε λίγες μέρες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής η θέση μας είναι σαφής. Πρέπει να διατηρήσουμε την απαγόρευση εμπορίου ελεφαντοστού. Υπάρχουν πολλές θέσεις από πλευράς των Αφρικανικών χωρών. Κάποιες προτείνουν να αρχίσει πάλι το εμπόριο αυτό, άλλες είναι κατά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής. Δεν θέλουμε το εμπόριο ελεφαντοστού να ξαναρχίσει. Το θέμα τώρα μπορεί σε ελεφάντων της Αφρικής. Είτε τους βάζετε στο πρώτο ή στο δεύτερο παράρτημα της ΙΤΕΣ, το πρώτο μιλάει για πλήρη απαγόρευση. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα στο ότι είμαστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης εμπορίου ελεφαντοστού το να βάλουμε στο παράρτημα 1 ή δύο τους ελέφαντες, αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την πλήρη απαγόρευση ελεφαντοστού. Ελπίζω να απάντησα έτσι στις ερωτήσεις σας. Τέλος. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο ρόλο των συμφωνιών ελεύθερων ε, συναλλαγών. Εδώ θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη χρήση των συμφωνιών αυτών και να χρησιμοποιούμε το εμπορικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες στο θέμα του, των καταλόγων με τα απειλούμενα είδη. Οπότε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ενισχύουμε και τις σχέσεις μας με τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων με τις μεταφορές ε, και άλλα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η συγγήτρια τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους για τη στήριξή σας στη γνωμοδότησή μου. Ελπίζω να μπορέσουμε πράγματι να ενισχύσουμε ε, τους ελέγχους και να αποτελέσουμε την προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πρότασή της που είναι πάρα πολύ σημαντική για να χτίσουμε εκεί απάνω. Ελπίζω τα σχόλια σας όντως να υλοποιηθούν στην ΣΥΤΕΣ. Εσείς λέτε ότι δεν έχει μεγάλη σημασία το σε ποιο παράρτημα θα μπουν οι ελέφαντες. Εμείς πιστεύουμε πως ναι αυτή η συγκεκριμένη στιγμή είναι η πιο κατάλληλη για να ε, καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Θα αναφερθώ εδώ σε δύο πράγματα. Θα πάω στο Johannesburg στη διάσκεψη αυτή της ΣΥΤΕΣ και όταν επανέλθω θα σας ενημερώσω φυσικά για τόσο θα έχουν διεξαχθεί εκεί και για τις συνομιλίες που θα έχω τότε. Πάντως, θέλω να σας υπενθυμίσω επικεντρώσετε στις τροπολογίες σας στο πρόγραμμα δράσης. Το Δεκέμβριο θα έχουμε και κάτι παραπάνω. Αύριο στις 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έμα. Ωραία. Τελειώσαμε αυτά. Αύριο στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τροπολογίες 26 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε εδώ, οπότε ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και σα ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα την εισηγήτρια. Τώρα φτάνουμε στο σημείο 23 στην ημερήσια διάταξη. Είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας. Θα δώσω λοιπόν... Μάλλον πρώτα θα σας πω ότι 1η Ιουλίου έχουμε μια επέτειο. Πέντε χρόνια ισχύει η συμφωνία αυτή. Ο κύριος Σάνφελτ από το ΕΛΚ έκανε την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας και δίνω και το λόγο αμέσως αυτόν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Λοιπόν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας, πέντε χρόνια πέρασαν από τότε, όπως αναφέρθηκε. Γι' αυτό προετοιμάζουμε αυτή την έκθεση, την οποία θα ήθελα να σας παρουσιάσω εδώ. Σήμερα έχουμε μόνο την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πρώτη συζήτηση. Η έκθεση θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο. Υπάρχει αρκετός χρόνος λοιπόν. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε ή τις προτάσεις σας, ε, τις απόψεις σας μπορείτε να μου τις αποστείλετε και μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μου προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα όμως ήδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη θετική συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αλλά επίσης ε, και τους συνεργάτες από τη Γραμματεία και από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Τους ευχαριστώ όλους λοιπόν. Τώρα οι λεπτομέρειες. Τις λεπτομέρειες θα σας τις παρουσιάσω τον Οκτώβριο με την έκθεση που θα καταθέσω όταν θα έρθει η χρονική στιγμή να συζητηθούν τα θέματα της έκθεσης. Σήμερα μόνο κάποιες γενικές πληροφορίες. Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε με την πρώτη συμφωνία της πρώτης γενεάς, έχουμε την πρώτη συμφωνία νέας γενεάς ενώπιών μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτού του είδους η συμφωνία νέας γενεάς, αυτού του είδους η συμφωνία νέας γενεάς είναι σημαντική υπόθεση. Είναι σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό κάθε πρίσμα η Κορέα, οπωσδήποτε Εμάς μας ενδιαφέρουν όμως κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και επιπτώσεις. Η Κορέα είναι για μας μια χώρα εταίρος, σε αυτό πρέπει να εστιαστούμε, χώρα εταίρος που όσον αφορά το επίπεδο της, του οικονομικού όγκου και των επενδύσεων είναι πολύ σημαντική. Η νέα μορφή συμφωνιών συναλλαγών, ελεύθερων συναλλαγών. Ξεκινά λοιπόν, ας το πω με την συμφωνία με την Κορέα σε αυτή τη φάση. Και η πείρα που έχουμε αποκομίσει από αυτές τις ε, πρώτες συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο και σε άλλες χρήσεις, προς άλλες κατευθύνσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, ποια θα είναι η τελική τους έκβαση, ποια θα είναι τα τελικά αποτελέσματα. Τι θα μπορούσαμε όμως μετά από πέντε χρόνια να πούμε, μετά από πέντε χρόνια εμπειρίας που έχουμε και πείρας που έχουμε συλλέξει. Έχουμε μπροστά μας μια επιτυχή ιστορία, μιας χώρας ε, με επιτυχίες. Οι ε, επιπτώσεις, οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας είναι θετικές ή και πολύ θετικές ε, κιόλας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τη δημοκρατία της Κορέας. Και εδώ ακριβώς θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια στοιχεία, σε, κάποια, σε κάποιους συντελεστές. Στη σύναψη της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, μετά τη σύναψη αυτή, αυξήθηκαν οι εξαγωγές ε, κατά 50% προς την Κορέα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 5% μόνο. Αλλά όπως θα αναφέρω υπήρξαν κάποιοι συντελεστές που εξηγούν αυτό το φαινόμενο, αυτή την μονοβαρή ε, κατάσταση πραγμάτων. Από πλευράς των Κορεατών έχουμε πολύ θετικές επιπτώσεις. Κατά το έτος 2015 είχαμε ρεκόρ που σημειώθηκε όσον αφορά το εμπόριο, τις εμπορικές συναλλαγές. Και όσον αφορά τον εμπορικό ισολογισμό, τον απολογισμό που μπορούμε να κάνουμε. Και οι εξαγωγές σε σχέση με την Κορέα όλο και αυξάνονται. Η συμφωνία αυτή αφορά όχι μόνο θέματα εμπορίου, αλλά και τις υπηρεσίες την παροχή υπηρεσιών και συγγνώμη επενδύσεις επίσης σίγουρα και τις επενδύσεις. Οι Κορεάτες ομόλογοι θέλουν το πρόβλημα των επενδύσεων να το τονίσουν πιο έντονα και να ληφθεί πιο έντονα υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Κορεατών και η Κορέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο όγδος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ακόμα και πριν από την προσυπογραφή της ε, συμφωνίας αυτής, υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες που είχαν τότε διατυπωθεί. Διατυπώθηκαν αμφιβολίες όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Τώρα, Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και αυτό το θέμα, υπήρξαν κάποιοι φόβοι όσον αφορά την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε σχέση με τις, ε, την κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτοί οι φόβοι όμως δεν ε, αποδείχθηκαν, δεν καταδείχθηκαν βάσιμοι, ήταν ασύστατοι και ο όγκος αυξήθηκε κατά 206% όσον αφορά τις εξαγωγές της Ένωσης ε, και οι εισαγωγές από την Κορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά 43% αυξημένες. Ακόμα και ο όγκος των υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε, διότι φυσικά έχουμε τα δικά μας σημεία αναφοράς και είναι σαφές αυτό. Άλλου είδους υπηρεσίες παρέχονται, για παράδειγμα, από εμάς, τους Ευρωπαίους, σε σχέση με τους Κορεάτες διαφορετικές, διαφορετικού τύπου υπηρεσίες. Τι μπορούμε να πούμε μετά από όλα αυτά. Μπορούμε να δούμε ότι αυτή η συμφωνία ε, ελευθέρου εμπορίου, ελευθέρων συναλλαγών είναι χρήσιμη, είναι υποφελής Οι εταίροι μας, πολιτικοί αφενός αλλά και επιχειρηματίες από την Κορέα, επιβεβαιώνουν αυτή την πτυχή. Κατά το παρελθόν είχαμε ένα έλλειμμα όσον αφορά το εμπόριο με την Κορέα. 7,5 δις ευρώ ήταν αυτό το έλλειμμα μας. Τώρα όμως έχουμε ένα πλεόνασμα. 7,3 δις είναι το πλεόνασμά μας τώρα. Εμπορικό μας πλεόνασμα έναντι των Κορεατών. Κατά το παρελθόν έλλειμμα 7,5 δις, τώρα πλεόνασμα 7,3 δις. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν να επεξηγήσουν το φαινόμενο αυτό. Οι πολιτικοί οι οποίοι είναι ε, υπεύθυνοι δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκλειστικά σε αυτούς οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Όμως παρόλα αυτά είναι σημαντική αυτή η πτυχή είχαμε μια πιο αποδυναμωμένη ε, τάση όσον αφορά τις ε, εισαγωγές. Ε, ίσως εδώ πρέπει να υπάρξουν οι σωστές επεξηγήσεις, τα σωστά συμπεράσματα για να μην καταλήξουμε σε λαθασμένες διαπιστώσεις. Επίσης, η κατάσταση που απορρέει και από την κρίση την οποία αντιμετώπισε η Ευρώπη και μάλιστα αρκετά χρόνια μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να ε, ξεφύγουν από αυτή την κρίση, να απελευθερωθούν από αυτή την κρίση. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η αύξηση των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων. Εδώ το ότι οι επενδύσεις αυτές αναφέρονται όχι μόνο στην Κορέα, αλλά και σε άλλες χώρες της, από Ανατολής, από, ε, ε, Ανατολικής Ασίας. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουν καταχωρηθεί ξεχωριστά τα κορεατικά εμπορεύματα ή αγαθά. Ίσως αυτό είναι μια εξήγηση για την αποδυνάμωση σε σχέση με τις τάσεις ε, που σημειώθηκαν. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και για διάφορους άλλους λόγους για την ανάπτυξη του εμπορίου μας συνολικά με την Κορέα. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή, την υλοποίηση των μέτρων για αυτή την εμπορική συμφωνία, πρέπει εδώ να αναφερθούν οι συμβουλευτικές ομάδες, εσωτερικές δομικές συμβουλευτικές ομάδες, διότι για τα κράτη-μέλη δεν πρέπει μόνο οικονομικά θέματα να είναι σημαντικά, αλλά και τα εργασιακά, τα θέματα των εργαζομένων και τα θέματα των πολιτικών ε, ελευθεριών. Συμφωνίες λοιπόν ελευθέρων συναλλαγών, ελευθέρου εμπορίου έχουν σήμερα μια μεγαλύτερη ε, εμβέλεια και σπουδαιότητα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά φυσικά και η κατάσταση των πολιτών, για παράδειγμα στην Ευρώπη και παγκόσμια, πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ε, εξεταστεί αντίστοιχα. Αυτό το στοιχείο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας. Αυτές οι πληροφορίες που σας παρουσίασα και σας, ε, ε, μόλις σας παρήχα, δεν σημαίνουν υποχρεωτικά ότι έχουμε μόνο θετικά φαινόμενα και, και, ε, μια θετική αποκλειστικά τάση. Γι' αυτό τον λόγο μετά από πέντε έτη όπως προβλέπετε υπάρχει και μια επανεξέταση, μια αναθεώρηση ώστε αν χρειαστεί να υπάρξουν ε, διορθωτικές κινήσεις, αντισταθμιστικές κινήσεις να δούμε τι χρειάζεται να γίνει από τους συμβαλόμενους εταίρους. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ρήτρα για τις άμεσες εξαγωγές και που τους παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που επισημαίνουν ότι φύσταται πρόβλημα σχετικά πρέπει να επανεξεταστεί και όσον αφορά την ε, ρήτρα για τις επισκευές η ευρωπαϊκή πλευρά θεωρεί ότι και τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας όπως copyright διαδραματίζουν ένα ρόλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και οι φυτοϊγειονομικές επίσης διατάξεις και ρήτρες και αυτές διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα που είναι σημαντικά για μας. Για παράδειγμα, τα πορτοκάλια για την Ισπανία ή το χείριο κρέας, για παράδειγμα, για την Πολωνία. Εδώ δεν έχουμε μόνο το θέμα των προσκομμάτων στο θεμητό εμπόριο, οι προσκόμματα και εμπόδια τα οποία αναφύονται, προβλήματα υφίστανται και παρουσιάζονται στις εμπορικές μας σχέσεις και με άλλους εταίρους μας, ε, ε, όπως εδώ και με τους Κορεάτες. Η κορεατική πλευρά αναφέρει το γεγονός ότι το ζήτημα των επενδύσεων έχει ένα ξεχωριστό ρόλο. Θέλω να διατυπώσω την εξής θέση. Έχουν δίκιο οι Κορεάτες σε αυτό που λένε, διότι αυτό το πρόβλημα στην αρχική συμφωνία δεν έτυχε σωστή αντιμετώπιση και δεν επιλήθηκε όπως έπρεπε. Υπήρχε ένας λόγος γι' αυτό. Στην αρχή δεν είχε εντολή, επαρκή εντολή η ευρωπαϊκή πλευρά ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα επαρκώς. Από την άλλη πλευρά η Κορέα είχε ξεχωριστές άλλες συμφωνίες για την προστασία αυτών των ε, ε, θεμάτων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν 23 τέτοιες ξεχωριστές συμφωνίες που έχει συνάψει η Κορέα. Και αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα για επιχειρήσεις που ε, ε, δραστηριοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Διότι πολλές φορές απορρέουν προβλήματα από αυτές τις διμερείς συμφωνίες και αυτό επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξελιχθεί, έχει, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα όσον αφορά την προστασία των ε, επενδύσεων. Διαφορετικά αντιμετωπίζονται οι επενδύσεις και η προστασία των επενδύσεων σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Και η ευρωπαϊκή και η κορεατική πλευρά θα πρέπει εξετάζοντας τα θέματα αυτής της συμφωνίας να εστιαστούν σε αυτό το ζήτημα. Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες διαδραματίζουν ένα ρόλο και πρέπει να λυθούν υπόψη. Επίσης κοινωνικά θέματα, κοινωνική, ε, κοινωνικά ζητήματα καταδεικνύουν ότι άξιζε τον κόπο να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Είναι λοιπόν θετικές οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα για την σύναψη περαιτέρω τέτοιων συμφωνιών με άλλα περαιτέρω κράτη-μέλη. Φυσικά Όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επιτήρησης ε, και παρακολούθησης και αν χρειαστούν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ή αντισταθμιστικές κινήσεις στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν. Υπήρξε θετική αντιμετώπιση στην Ευρώπη. Οι εκπρόσωποι διαφορετικών τομέων τοποθετήθηκαν και στην Ευρώπη αλλά και στην Κορέα και με θετικό πνεύμα. Και πιστεύω τούτων λεχθέντων ότι στην έκθεση που θα σας παρουσιάσω θα υπάρξουν επαρκώς τα θεμέλια ώστε να κριθεί με θετικό πνεύμα αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στους και ηγητές. Ο κύριος Σούστερ από τους ε, σοσιαλιστές. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση με την οποία συμφωνώ σε πολλά σημεία. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχή συμφωνία αυτή που έχουμε ενώπιόν μας και μπορεί σίγουρα σε πολλά, σε πολλά θέματα να θεωρηθεί υποδειγματική. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η πολιτική στη Νότια Κορέα δεν κρίνεται πάντα με τόσο θετικό πνεύμα, διότι υπό το κορεατικό πρίσμα είναι ήδη μια δυσχέρεια το ότι υπάρχει, υπήρχε αυτό το έλλειμμα το οποίο επιβάρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από πέντε χρόνια και που έχει αναστραφεί πλήρως τώρα σε πλεόνασμα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται έτσι χωρίς αντιρρήσεις δεκτό. Υπάρχουν επικρίσεις για αυτή την κατάσταση πραγμάτων από την Κορέα. Συμφωνώ όμω ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ξεφύγει από την κρίση πολυσχηδός σε σχέση και με ε, ευρωπαϊκά κράτη και δείχνει αυτό ότι η αηφορία για την ανάπτυξη στην οικονομική πολιτική που ακολουθούμε όχι μόνο οικονομικά δημιου... μας θέτει προβλήματα αλλά και στο... επιβαρύνεται πολλές φορές λόγω αυτής της κατάστασης και το εξωτερικό εμπόριο και πρέπει να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις σε συμφωνία πάντα με τους Κορεάτες διότι το τελικό, η τελική έκβαση όλων αυτών πρέπει να είναι και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας να αυξηθεί η εμπορική δραστηριότητα αμφωτέρωθεν. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και συναποτελούν μια σημαντική μεταβολή των πραγμάτων και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αφενός το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα κίνητρα των Κορεατών επικεντρώνονται ε, συγκεκριμένα στο, λόγο, στο θέμα το ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία προστασίας επενδύσεων με όλα τα κράτη-μέλη όπου θα έχουν δικαιώματα οι επιχειρήσεις της Κορέας να ασκήσουν προσφυγές ε, ε, ή να διεκδικήσουν δικαιώματα αν υπάρχουν αλλαγές ή μεταβολές όμως οι νόμιμες ε, νομικές μεταβολές και νομοθετικές μεταβολές δεν μπορούν να αποτελούν λόγο να ε, θεωρηθεί κάτι καταχρηστικό. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε όπου από την ευρωπαϊκή πλευρά δεν έχουμε κλασικά συστήματα SDS, δηλαδή συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, αλλά η λύση μπορεί να καταλήξει μόνο υπό τη μορφή ενός ε, ε, διεθνούς ε, διαιτητικού φορέα ή δικαστηρίου που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη θα διατηρήσουν το δικαίωμα νομοθετικών αλλαγών και προσαρμογών χωρίς περιορισμούς, μια και είναι κυριαρχικό τους δικαίωμα αυτό. Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό υπό το πρίσμα μας είναι ότι η Νότια Κορέα δεν έχει πλήρως προσαρμοστεί και δεν τηρεί πλήρως όλες τις πτυχές της συμφωνίας. Για παράδειγμα, σε σχέση με κυριαρχικά δικαιώματα εργατικά των εργαζομένων, πρέπει πολλά να γίνουν. Υπάρχουν εδώ υπό πολλές αμφισβητήσεις, ε, ε, συλλήψεις ε, συνδικαλιστών και που όχι μόνο απειλήθηκαν αλλά και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για μας. Το χαιρετίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτό το ζήτημα. Εμείς θα θέλαμε να πάμε λίγο πιο πέρα η επίλυση, η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και η διασφάλιση των θεμελιωδών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Νότια Κορέα είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη σχέση μας με την Νότια Κορέα. Πρέπει να έχουν ε, ίδιο βάρος και αξία οι σχέσεις ε, για τα εργασιακά και τα εργασιακά θέματα όπως τα άλλα σε σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Δεν μπορούμε εδώ να παραβλέψουμε αυτό το θέμα στο τέλος εκτιμώντας τα πράγματα σωστά νομίζω ότι ήταν μια επιτυχής έκβαση αυτή η συμφωνία και για τις δύο πλευρές και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει επικοδομητικά να προχωρήσουμε ευχαριστώ ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάποτα από το ΕΣΥΑΡ e τώρα έχει το λόγο. Μάλιστα, συμφωνώ με τον εισηγητή. Η συμφωνία με την Κορέα είναι μια επιτυχία. Όπως κάθε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης που είναι θετικό. Πρέπει εδώ σε σχέση με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα με την Νότια Κορέα να μεριμνήσουμε να, να τηρούνται, να είναι σεβαστά. Εδώ μία παρατήρηση θα ήθελα ως οικονομολόγος σε σχέση με τα πλεονάσματα, τα εμπορικά πλεονάσματα να κάνω. Είναι ικανοποιητικό φυσικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα έχει από ένα μια επιβάρυνση του παρελθόντος τη μετέφερε αυτήν σε ένα πλεόνασμα ε, την υπερχρέωση που είχε. Και τώρα οι Κορεάτες θα πρέπει σε σχέση με την, ε, το κράτος ε, δικαίου στην Κορέα να μεριμνήσουμε και να δούμε πώς ε, αυτό το πλεόνασμα εξηγείται και σε τι βασίζεται. Αν βρίσκονται, για παράδειγμα, αγαθά τα οποία όλο και περισσότερο εξάγονται προς την Κορέα, τότε αυτό θα αυξήσει την παραγωγικότητα των Κορεατών είναι λοιπόν μια προσωρινή θα λέγαμε, ένα προσωρινό φαινόμενο αυτό το πλεόνασμα και θα πρέπει να δούμε την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των Κορεατών και παραγωγικότητα που ίσως θα μπορούσε να ε, μεταβάλει πάλι τα πράγματα. Σε σχέση με το πλεόνασμα το οποίο ε, έχει τώρα ε, δημιουργηθεί ενώ πριν είχαμε μια ελληματική κατάσταση για την Ευρώπη πρέπει να οδηγήσει σε, μια, ένα κέρδος και για το εμπόριο οικονομικό αλλά και για την ευημερία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο για την Άλντε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Αλεξάνδερ Λάμστορφ είναι εκείνος ο οποίος ε, θα ήταν αρμόδιος, μια και όμως δεν παρίσταται, θα μπορούσα να αναφέρω εγώ κάποια πράγματα εξ ονόματός του. Όχι οτιδήποτε, αλλά ίσως ε, δύο-τρία πράγματα. Είχα και εγώ τη δυνατότητα να συμμετάσχω από πλευράς μου στην αποστολή μας στην Κορέα, Νότια Κορέα. Και βλέπει κανείς ότι πρόκειται για μια επιτυχή συμφωνία αλλά υπάρχουν επίμαχα θέματα όσον αφορά τα συνδικάτα και φυσικά οι εργασίες που διεξάγονται από πλευράς μας διεξάγονται με βάση τις δικές μας αξίες και αρχές και πρέπει να δούμε πώς οι άλλοι αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα αξιακά. Όταν σημαίνει πλεόνασμα για την Ευρώπη αυτή η συμφωνία Κάποιοι Ευρωπαίοι ανέφεραν όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία ότι υφίστανται προβλήματα, είπαν. Όμως οι Νοτιοκορεάτες προσπαθούν τις δικές τους μάρκες και τα δικά τους προϊόντα να ευνοήσουν και εδώ υπάρχει η άποψη ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα τα ευρωπαϊκά οχήματα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα όπως τα κορεατικά. Και εδώ ίσως υπάρχει λοιπόν ανάγκη για βελτιώσεις αλλά όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για μια καλή συμφωνία για μας τους Ευρωπαίους. Ίσως υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, ένα ερωτηματικό για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, για το intellectual property rights και το copyright. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα ξαναδούμε και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ώστε οι Κορεάτες από πλευράς τους να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εναντί των Ευρωπαίων και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των καλλιτεχνών, των μουσικών και των, ε, της προστασίας του έργου τους. Σε σχέση με την συζήτηση αυτή, με κάποιες προσθήκες λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις, διευρύνεται το πλαίσιο το οποίο εξετάζουμε. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή για τα στοιχεία που μας έδωσε και την άποψή του για την επιτυχημένη ιστορία και την ανάπτυξη της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Ε, πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως ιστορία επιτυχίας ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θυμάμαι και τα τελευταία είχε πει ο κύριος δεμάτη ε, ε, ο οποίος πάντα πιστεύει ότι πρέπει να υποχράβουμε περισσότερες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και η Κορέα είναι το χαρτί της επιτυχίας για κάτι τέτοιο. Παρά τα θετικά στοιχεία βέβαια, Υπάρχουν κάποια στοιχεία, παραδείγματο χάρη για τον ευρωπαϊκό ε, τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία, στη χώρα μου για παράδειγμα, ή κάποια είδη πολιτεολία τα οποία εισάγονταν από την Ιαπωνία και ίσως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βάλει κάποιο όριο, να δει λίγο και πίσω από τις αδρές γραμμές πρέπει να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση αυτής της συμφωνίας, όχι μόνο με ορίζοντα πέντε ετών, αλλά να δούμε και την εφαρμογή και τις συνέπειες που υπάρχουν για την γενική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των χωρών μας ε, μακροπρόθεσμα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη ομάδα παρακολούθησης ε, να συνοδεύει την ε, περαιτέρω εφαρμογή αυτή της συμφωνίας και τι συνέπειε έχει αυτή για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην οικονομία και με τη διαφορά που υπάρχει με την οικονομία της Κορέας. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της αναφέρει ότι ότι από τα 11 χρόνια πλεονασμάτων που έχουμε ε, στο εμπόριο Κορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να θεωρείται μόνο ε, αποτέλεσμα της ε, ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών αλλά και ε, λόγω άλλων αλλαγών. Μήπως δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τα στοιχεία αλλά να εξετάσουμε λίγο πιο ε, στενά που υπάρχει αύξηση, που υπάρχει ανάπτυξη, που υπάρχει μείωση αν σχετίζονται με τις οικονομικές εξελίξεις και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, το ισοζύγιο πληρωμών, τι σχέση έχει οι συναλλαγματικέ ισοτιμίες επίση. Επομένως, θεωρώ ότι θα πρέπει να κρίνουμε τις συνέπειες αυτών των συμφωνιών και εν ώψη της ε, συνόδου του G20 που θα ασχοληθεί με την παγκόσμια οικονομία, το οικονομικό και διεθνές εμπόριο και τις ε, διεθνείς εξελίξεις. Ε, φαίνεται να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα πρέπει να να τα λαμβάνουμε υπόψη αυτά στις διαπραγματεύσεις μας σε πολυμερές, διμερές επίπεδο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι αν αλλάξει η ισοτιμία του ευρώ, θα έχουμε και πάλι μια χώρα η οποία δεν έχει κυρώσει τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Το είπε και ο κύριος Σούστερ βεβαίως αυτό. Υπάρχει και ντάμπινγκ εδώ, γι' αυτό και λοιπόν ζητάμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή της για την νέα νομοθεσία που έχει περάσει η χώρα, που δεν ε, βολτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες. Αντιθέτως, ε, η κατάσταση για κάποιες ομάδες ε, του εργατικό δυναμικού επιδεινώθηκε. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε ελεύθερο εμπόριο και εμπόριο για όλους και όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, η GUNGL επιμένει ότι θα πρέπει Όπως αναφέρεται και στην ε, ε, γνωμοδότηση Επιτροπής Απασχόλησης ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και ευκαιρία για να ζητήσουμε από την Κορέα να κυρώσει και να υπογράψει όλες τις ε, συμφωνίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις σχετικές συμβάσεις και να είναι αυτό υπό όρους για τη συνέχεια της ε, ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Συναλλαγών, ε, την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, δικαιώματα γυναικών εργαζομένων και παιδικής εργασίας. Και επομένω να μην υπάρχουν διακρίσεις και να γίνεται σεβαστή η αξιοπρεπής εργασίας. Θεωρώ ότι όλα αυτά ανήκουν στην πλήρη ανάλυση του αντικτύπου που έχει η εφαρμογή αυτή της ε, συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Κορέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Ο κύριος Δεκοντέη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα θετικά τους ε, σχόλια. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, 1η Ιουλίου είχαμε την 10 η επέτειο εφαρμογής της Συμφωνίας Ελευθέρου Συναλλαγών και τον περασμένο Δεκέμβριο η Συμφωνία ε, τέθηκε επισήμως ε, εν, ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης. Χαίρομαι που η Σογητή υπενθύμησε ότι αυτή η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου ε, είναι μια επιτυχημένη ιστορία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εσεί πολύ σωστά υπενθυμίσατε το πλεόνασμα και τα ποσοστά και την αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών που διαπιστώσαμε και που επιβεβαιώνουν το γεγονό ότι πρόκειται για επιτυχία. Τον Ιούνιο δημοσιεύθηκε ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρω Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας που περιλαμβάνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για τα εμπορικά μεγέθη ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέα. και φυσικά η έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Αναφέρθηκαν αρκετά στοιχεία σε κάποιε από τι ερωτήσει και θα ήθελα να σταθώ σε αυτά. Καταρχά, σαφώ και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης μέσω μιας δέσμης ε, τροποποιητικών μέτρων και ήδη συζητούμε με την κορεατική πλευρά τα συγκεκριμένα σημεία, ε, κυρίως ε, στην τελευταία Επιτροπή Εμπορίου τη Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κορέας. Η Επίτροπος ε, Μάλστρομ και ο εταίρος της από πλευράς Κορέας άρχισαν να συζητούν αυτή τη δέσμη των τροπολογιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ευαισθησίες και τα συμφέροντα της κάθε πλευράς. Η Κορέα προ το παρόν έχει επιδείξει θετική στάση για τη διαπραγμάτευση αυτή της δέσμη τροπολογιών με φυσικά κάποιες πολιτικές επιφυλάξει, οι οποίες συνδέονται και στην έλλειψη ισορροπία ή ε, την... Ε, ε, αντίληψη ότι ίσω είναι άνισε τα ωφέλη υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μας είπαν και το συζητούμε. Ε, θεωρούμε ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μπορεί να είναι επιτυχής αν υπάρχει μια ισορροπημένη ε, στάση και ε, ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Όπως πολύ σωστά υπενθυμίσετε, πρόκειται για μια διαπραγμάτευση κυρίως ενός κεφαλαίου επενδύσεων στη συμφωνία. Πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι επενδύσεις δεν αποτελούσαν τμήμα της ε, αποκλειστικής εμπορικής μας ερμοδιότητας και της εντολής μας. Επομένως, γι' αυτό και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία ε, με την Κορέα. Οι Κορεάτες μας εξήγησαν ότι δεν έχουν κάποια ανησυχία για τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επενδύσεις σε σχέση με τις ε, υφιστάμενες επενδυτικές συμφωνίες που υπάρχουν διμερώς και ε, υποστηρίζουν τους κανόνες προστασίας που θέλουμε να συμφωνήσουμε μαζί τους. Η μόνη ίσως ε, δυσκολία που πρέπει να συζητήσουμε ακόμα είναι ε, ο νέος μηχανισμός ε, επίλυσης διμερών διαφορών, το λεγόμενο σύστημα διαιτησίας, διότι οι Κορεάτες μας επεσήμεναν ότι δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί και δεν θα ήθελαν να είναι απαραίτητο η πρώτη χώρα που θα το θέσει υποδοκιμασία και επίσης επειδή ε, εξετάζουν και την, ε, ε, το ενδεχόμενο να ενταχθούν στην TPP που έχει τελείως διαφορετικό σύστημα επίλυσης διαφορεών από το ISDS και ομοιάζει αυτό το οποίο έχουν στις δικές τους ε, διμερείς συμφωνίες και άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ε, τους φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να πείσουν την Εθνική Συνέλευση της Κορέας ε, για το νέο σύστημα που προσπαθεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν ακόμα κάποιο κενό στο επενδυτικό κεφάλαιο, προσπαθούμε να τους πείσουμε, τους είπαμε ότι δεν θα ε, ξεφύγουμε από αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω συζητήσεις και εξηγήσει για το συγκεκριμένο σημείο. Γίνονται επίσης κάποιες συζητήσεις και για άλλα στοιχεία της δέσμης ε, τροπολογιών. Επειδή υπάρχουν ε, καλά στοιχεία, είναι περιορισμένα τα σχόλια για από τις δύο πλευρές. Στη Σεούλ στο Μάιο συναντήθηκαν ε, σε επίπεδο διευθυντών ε, υπεύθυνοι και θα γίνει άλλη μια συνάντηση ε, το Σεπτέμβριο εδώ στις Βρυξέλλες για να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Επίσης, έγιναν κάποια σχόλια για την αξιολόγηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών και όπως γνωρίζετε έχει ξεκινήσει με μελέτη για να αξιολογήσουμε την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Υπεγράφει τώρα μια συμφωνία με την επιχείρηση που έχει αναλάβει την ε, εκπόνηση της μελέτης στη Γερμανία και ελπίζουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τον Αύγουστο του 2017. Θα εξετάσουμε τα ωφέλη της συμφωνίας, θα εξετάσουμε απασχόληση, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, θα είναι πλήρης. Και ε, θα ενημερώνουμε τακτικά και την ιστοσελίδα με τα διάφορα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από την ε, εταιρεία που έχει αναλάβει και όταν θα λαμβάνουμε τα στοιχεία με τα χαράς να τα διαβιβάσουμε και σε εσά. Όσον αφορά το θέμα των συνδικάτων, το εργατικό δίκαιο και τη διεθνή ε, οργάνωση εργασίας, ε, αυτή είναι μία από τις ανησυχίες που έχουμε πράγματι και πολύ προσακτικά παρακολουθούμε την κατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων στην Κορέα. Όπως γνωρίζετε, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναγαρών παρέχει ένα θεσμικό μηχανισμό για να συζητούνται ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτει και τα εργατικά δικαιώματα. Στην τελευταία συνεδρίαση που έγινε λοιπόν για εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη, ε, ζητήσαμε από την Κορέα να λάβει μέτρα προκειμένου να κυρώσει όλες τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπως προβλέπονται από τη Συμφωνία Ελευθέρων Συνολαγών και σε μια κοινή δήλωση η Κορέα δεσμεύτηκε να μας δώσει πληροφορίες για το τι συγκεκριμένα βήματα έχει αναλάβει προκειμένου να το υλοποιήσει. Ε, θα το παρακολουθούμε λοιπόν, θα επανέλθουμε στη συζήτηση, κυρίως στην επόμενη Επιτροπή Εμπορίου που θέλουμε να ε, διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Μαζί με τις κορεατικές αρχές ε, η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία ξεκίνησε ένα ε, σχέδιο εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή της Σύμβασης ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθμός 111 για, την, για τις διακρίσεις. Επομένως, ε, ε, σας διαβεβαιώ ότι ο Επίτροπος Μάλστρομ παρακολουθεί στενά το θέμα. Κάτι επιπλέον τώρα για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και τα λεγόμενα δικαιώματα δημόσιων ε, παραστάσεων. Η Κορέα δεν συμμορφούνται πλήρω με τις διεθνείς υποχρεώσεις για αυτά τα δικαιώματα και επομένως τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία Ελευθέρων Συνολογών Ευρωπαϊκή Ένωση Κορέα, Θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία για να προχωρήσει η διαδικασία συμμόρφωσης. Ε, για αρκετά χρόνια είχε σταματήσει αυτό στην ε, ε, Κορεατική Εθνοσυνέλευση από Κορεάτες βουλευτέ. Το Μάρτιο Φέτο πέρασε επιτέλους το νομοσχέδιο από την Εθνοσυνέλευση, αλλά δυστυχώ η διατύπωση ήταν κάπω πιο ήπια και επομένω η αναθεωρημένη πράξη δεν αντιμετωπίζει πλήρως τις ανησυχίες ε, των κατόχων πραγματικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βελτιωθεί η κατάσταση είμαστε τώρα στη διαδικασία ε, εξέτασης των λεπτομαριών που χρειαζόμαστε στη λεγόμενη ε, δευτερογενή νομοθεσία που θα προκύψει από αυτό και παρακολουθούμε το θέμα στενά και με τον αρμόδιο κλάδο και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με την αντιπροσωπεία και τα κράτη-μέλη στην Κορέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στον εισηγητή μας τώρα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ φυσικά όλους που παρενέβησαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους. Οι θέσεις ε, που παρουσίασα από πλευράς μου στις παρεμβάσεις που ακούστηκαν επιβεβαιώθηκαν. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω αυτό το οποίο ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα που αναφέρεται και στην έκθεσή μου εξάλλου Δηλαδή, οι πνευματικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να είναι σεβαστά εργασιακά δικαιώματα και αυτό το έλαβα υπόψη. Αυτή τη συμφωνία την αξιολόγησα εγώ με βάση τις οικονομολογικές μου γνώσεις ως επιστήμον, ως επιστήμον και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας, ποσοτικά αποτελέσματα, δεν είναι μόνο κάτι που αφορά άμεσα το άμεσο εμπόριο, αλλά και την οικονομία διαφορετικών χωρών. Διότι εδώ έχουμε πολλούς συντελέστες και παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών και η οικονομική κατάσταση παγκόσμια και αυτή διαδραματίζει ένα ρόλο. Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ένα πράγμα, ότι οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας μπορούν να χαρακτηριστούν θετικές, αδιαμφισβήτητα. Υπάρχει μια ασάφεια όσον αφορά τις διαστάσεις, των, το εύρος αυτών των θετικών επιπτώσεων. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την εξωτερική αξιολόγηση και ανάλυση, πράγμα που ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η ανάλυση δεν θα πρέπει μόνο οικονομικούς συνταλεστές και παράγοντες να λαμβάνει υπόψη, αλλά και κοινωνικά στοιχεία, πολιτιστικά, θέματα τα οποία συνεπηρεάζουν την κατάσταση γενικά και που θα πρέπει και μελλοντικά να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τα συνδικάτα και τα δικαιώματά τους. Όσον αφορά τον σεβασμό και το, τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ε, της ILO μας ενδιαφέρει άμεσα το θέμα όπως και τα άλλα μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ γι' αυτό αυτά τα θέματα υπήρξαν κάποιες συναντήσεις που διεξήχθησαν ήδη με τους εκπροσώπους των κορεατικών συνδικάτων και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων της Κορέας. Είχαμε επίσης επαφές με κορεάτες πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από την Νότια Κορέα. Και κατά τα άλλα επισημάναμε και αναφέραμε ότι όλα αυτά τα θέματα θα είναι πολύ σημαντικά για μας σε σχέση με την αξιολόγηση στην οποία θα προβούμε αυτής της συμφωνίας και αν θα χρειαστεί για ενδεχόμενα κιόλας να τροποποιηθεί το κείμενο αυτής της συμφωνίας ε, οι διατυπώσεις μελλοντικά. Αυτές οι προσδοκίες λοιπόν που αναφέρθηκαν σίγουρα θα υλοποιηθούν, σίγουρα θα γίνουν αυτά. Και μια άλλη σκέψη που θα ήθελα από πλευράς μου να λάβετε υπόψη όσον αφορά το προηγούμενο θέμα στο οποίο ε, εστιαστήκαμε. Επρόκειτο για το εμπόριο με την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Φαίνεται φαινομενικά να είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα αποξενωμένο από το θέμα που συζητούμε. Όμως υπάρχει μια διασύνδεση εδώ Κάναμε λόγο χθε για τις συμφωνίες μεταξύ, εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Αφρικής για παράδειγμα. Πρόκειται ακριβώς για το επίπεδο ευημερίας και διαβίωσης ε, των ανθρώπων, την καταπολέμηση της φτώχειας, ε, την προώθηση, προαγωγή της ευημερίας, ε, τις καλύτερες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να διασφαλίζεται η γνώση, είναι το μεγαλύτερο εργαλείο, το καλύτερο εργαλείο για να καταπολεμηθεί αυτή η παθολογία και αυτά τα παθολογικά συμπτώματα που παρουσιάζονται. Δεν μπορεί να επιτευχθεί πολιτισμική και πολιτιστική πρόοδος ε, εκτός Ευρώπης χωρίς ε, την οικονομική ε, ανάπτυξη ως συντελεστή που θα επηρεάζει τα πράγματα και τις καταστάσεις. Συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών και εμπορίου είναι πολύ σημαντική συνιστόσα ως προς αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Τον Οκτώβριο θα συζητήσουμε στις 12 και 13 Οκτωβρίου πάλι. Το χρονοδιάγραμμα θα διευκρινιστεί παρετέρω πιο συγκεκριμένα τη συνέχεια. Είμαστε στο σημείο 24. Διάφορα. Εγώ δεν έχω διάφορα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για το έργο σας και ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους, τη γραμματεία κλπ. Λίγη συνεδρίαση.